δημοσιευτούν στα κείμενα που ευτήθηκαν σε αυτή τη σύνοδο μαζί με τα ονόματα όσων έχουν υπογράψει το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 17 ε, Ιουνίου 2010. Καλωσορίζω λοιπόν τον ε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σας καλωσορίζω κύριε. Πριν περάσουμε στην ε, συζήτηση θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Χερμάν Φαναρομπό, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή ήταν η πρώτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από όταν έγινα πρόεδρος, η οποία δεν είχε ως αντικείμενο κατεπήγοντα γεγονότα. Ήταν μια κανονική συνεδρίαση και οι αποφάσεις που λάβαμε είχαν μεγάλη σημασία ειδικά σε σχέση με την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης και το τι θα κάνουμε πέρα από την κρίση και πώς θα βελτιώσουμε τη μακροπρόθεσμη οικονομική απόδοση της Ευρώπης. Πρόσφατα επιδείξαμε ισχυρή πολιτική αποφασιστικότητα για την διασφάλιση της σταθερότητας του ευρώ. Χάρηκα που σε αυτή τη συνεδρίαση είδα παρόμοια αποφασιστικότητα για να ενισχυθεί η μακροπρόθεσμη οικονομική μας ισχύς για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για δουλειές και ανάπτυξη συμπεριλαμβανόμενη στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020. Βασιζόμενη στη δουλειά της Κομισιόν και των Συμβουλίων εγκρίναμε τους πέντε κύριους στόχους τους οποίους γνωρίζετε και τους οποίους θεωρούμε κρίσιμους για να αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης, που είναι ουσιαστικός εάν είναι να διατηρήσουμε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής με έναν πληθυσμό ο οποίος γυράσκει και να παραμείνουμε ένα παίκτη στην παγκόσμια σκηνή. Γνωρίζω πως κάποιοι σε αυτή την αίθουσα και αλλού έχουν εκφράσει εμφιβολίες και αναρτήθηκαν εάν η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 έχει καλύτερα αποτελέσματα από την προηγούμενη στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία γενικά θεωρείται ανεπαρκής. Είναι πεποίθησή μου πως πράγματι μπορεί. Εσκεμένα εστιάσαμε σε λίγους στόχους, αντί για πληθώρα στόχων που χάθηκαν στη στρατηγική της Λισαβόνας. Είναι ζωτικοί στόχοι και ενσωματώνουν την κοινωνική, περιβαλλοντική και εκπαιδευτική διάσταση που, στις οποίες σωστά επέμεινε το Κοινοβούλιο. Θα εστιάσουμε συνεχώς σε αυτούς τους ε, στόχους και θα έχουμε ετήσιες αναθεωρήσεις. Θα έχουμε εθνική ανάλυση του κάθε στόχου και όχι μόνο ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Οπότε θα έχουμε ρεαλιστικά μέτρα για να δούμε πώς είναι η αποδοσή της κάθε χώρας. Πάνω απ' όλα προσπάθησα η διαδικασία να θεωρηθεί ότι είναι κάτι που ανήκει στα καράτη-μέλη έτσι ώστε να μην το θεωρούν ως κάτι που υιοθετήθηκε στις Βρυξέλλες και μετά να το αγνοήσουν. Αλλά να το θεωρήσουν κάτι το οποίο είναι κομμάτι αναπόσπαστο της εσωτερικής τους οικονομικής στρατηγικής. Βασίζομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συνεχίσει να ασκεί πίεση για την εφαρμογή της στρατηγικής για το 2020. Πρέπει να η αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα του πώς αξιολογούμε την κατάσταση της Ένωσής μας. Χάρηκα για το ότι όταν εσείς κύριε Πρόεδρε απευθυνθήκατε στους αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων στην ε, αρχή της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα επισημάνατε πως το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τη στρατηγική του 2020. Αυτό ήταν ευπρόσδεκτο. Ταυτόχρονα γνωρίζω πως υπάρχουν κάποιοι, εδώ σε έσως και αλλού, που ανησυχούν για την μέθοδο που χρησιμοποιείται για να εφαρμοστεί η στρατηγική. Μήπως είναι, όπως κάποιοι είπαν, πάρα πολύ διακυβερνητική μέθοδος εργασίας. Θα επισημάνω απλώ πως η βελτίωση της οικονομικής απόδοσης της Ευρώπης απαιτεί την χρήση μιας σειράς μέσων. Κάποια από αυτά είναι εθνική αρμοδιότητα, άλλα είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε και υιοθετούμε κοινή νομοθεσία για την κοινή μας αγορά, για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, για την πολιτική ανταγωνισμού, για το εμπόριο, την προστασία των καταναλωτών και για άλλα ζητήματα. Επίσης, χρησιμοποιούμε τον προπολογισμό της Ένωσης, ειδικά τα διαρθρωτικά ταμεία και τα προγράμματα έρευνας. Σε όλα αυτά, ο ρόλος της Κομισιόν είναι κέριος. Αλλά βασικές πτυχές της οικονομικής μας απόδοσης παραμένουν εθνική αρμοδιότητα, μεταξύ των οποίων και η εκπαίδευση αν είναι να είμαστε επιτυχείς πρέπει να κινητοποιήσουμε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης σε μια κοινή προσπάθεια. Σύμφωνα με τη συνθήκη, και αναφέρω τώρα το άρθρο 121, τα κράτη-μέλη θα θεωρούν τις οικονομικές πολιτικές ζήτημα κοινή ανησυχίας και θα τις συντονίζουν εντός του Συμβουλίου. Ο συντονισμός αυτός θα βασίζεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και περιλαμβάνει όλα τα θεσμικά όργανα με συνεισφορά και της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου και αυξάνουμε το εύρος αυτού του συντονισμού όπως ακριβώς αυξάνουμε και το εύρος του τι κάνουμε με την ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως παραδείγματος χάρη στον τραπεζικό τομέα. Και ο συντονισμό των εθνικών πολιτικών και η κοινή δράση στο επίπεδο της Ένωσης απαιτούνται. Το καθήκον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθώς φέρνει σε επαφή και τον πρόεδρο της Κομισιόν και τους αρχηγούς των κυβερνήσεων είναι να ορίσει κατευθυντήρες γραμμές και πολιτικές κατευθύνσεις και για τα δύο αυτά στοιχεία. Όσοι προσπαθούν να φέρουν σε αντιπαράθεση Κομισιόν και κράτη-μέλη δεν εξυπηρετούν την Ένωση. Θα ήθελα να προσθέσω πως είναι κάπως εύκολο να εξισώνουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με την διακυβερνητική μέθοδο. Είναι πλέον ένα θεσμικό όργανο της Ένωσης, λειτουργεί στο πλαίσιο της ισορροπημένης αρχιτεκτονικής της Ένωσης, όπως περιγράφεται στις συνθήκες. Συμπεριλαμβάνει ως μέλος τον πρόεδρο της Κομισιόν και τώρα έχει ως πρόεδρο κάποιον ο οποίος εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Ένωσης συνολικά και δεν εκπροσωπεί ταυτόχρονα μια εθνική κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα πρέπει να υποθέτουμε πως οι αρχηγοί κυβερνήσεων δεν είναι ικανοί να αντιληφθούν το ευρύτερο κοινό συμφέρον ή ότι δεν γνωρίζουν το ότι το εθνικό του συμφέρον είναι να έχουν μια ένωση η οποία λειτουργεί σωστά. Για να επανέλθουμε στη συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε και μια απόφαση η οποία κατά την άποψή μου έχει εξίσου μεγάλη σημασία με τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Ήταν η απόφαση να συσταθεί ένας πίνακας βαθμολογίας και ένα σύστημα επιτήρησης για να αξιολογήσουμε την ανταγωνιστικότητα και τις ανισορροπίες για να ανοιχνεύουμε νωρίτερα ανισορροπίες και επικίνδυνες τάσεις. Αυτές οι ανισορροπίες δεν τις είχαμε προσέξει στο παρελθόν, κυρίως γιατί δεν ορίζονταν στη συνθήκη ως ένα από τα κριτήρια του Μάστριχτ. Όμως έχουν ζωτική σημασία. Μάλιστα, η κατάσταση που αντιμετωπίζουν τώρα κάποια κράτη-μέλη έχει ως αιτία αυτές τις ανισορροπίες. Το ευρώ ήταν θύμα της ίδιας του της επιτυχίας. Ξεχάσαμε πως το κοινό νόμισμα χρειάζεται σύγκληση και μεταρρυθμίσεις. Λάθη έγιναν σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης τα τελευταία δέκα χρόνια, ας είμαστε ειλικρινείς, είναι συλλογική ευθύνη. Όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα, προτεραιότητά μας είναι να έχουμε ένα στιβαρό και υγιές τραπεζικό σύστημα. Ζητήσαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Ακοφή να υιοθετήσουν γρήγορα τις νομοθετικές προτάσεις για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και οι τρεις εποπτικές αρχές να μπορούν να ξεκινήσουν να δουλεύουν το 2011. Η συνεισφορά σας είναι ζωτική και η ευθύνη σας μεγάλη. Επίσης συμφωνήσαμε πως τα τεστ κοπόσεως των τραπεζών θα δημοσιευτούν το αργότερο το δεύτερο μισό του Ιουλίου. Ζητήσαμε από την Κομισιόν να κάνει γρήγορα προτάσεις για τις ακάλυπτες πωλήσει και τα ασφαλιστρά ομολόγων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε πως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εισαγάγουν ένα σύστημα εισφορών και φόρων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και συμφωνήσαμε να εξερευνήσουμε με τους εταίρους μας, τους G20, την δυνατότητα φόρου παγκοσμίω στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Μάλιστα συμφωνήσαμε σε μια κοινή θέση, σε μια σειρά ζήτημάτων που θα μας απασχολήσουν στην σύνοδο του Τορόντο τον G20 όπου εγώ και ο κύριος Μπαρόσο θα εκπροσωπήσουμε την Ένωση. Επίσης επαναβεβαιώσαμε την θέση μας για την επίτευξη των στόχων των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και συγκεκριμένα μέχρι το 2015 να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους παρά την οικονομική κρίση και να προχωρήσουμε περαιτέρω στην κλιματική αλλαγή. Συμφωνήσαμε υπό όρους να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ένταξης της Ισλανδίας και ε, καλωσορίσαμε την ε, αίτηση της Εστονίας να μπει στην ζώνη του ευρώ και τα δύο αυτά σημεία αποτελούν ένδειξη εμπιστοσύνη στην Ένωσή μα. Επίση, υιοθετήσαμε μια δήλωση για το Ιράν που τονίζει τις βαθύτερες ανησυχίες μας για το πυρηνικό του πρόγραμμα και ζητήσαμε από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών να υιοθετήσει μέτρα για να εφαρμοστούν οι κυρώσεις του ΟΗΕ και να συνοδευτούν απεραιτέρω μέτρα. Αποδεικνύουμε έτσι πως η Ένωση μπορεί να έχει κοινή θέση σε ένα από τα πιο λεπτά ζητήματα στην παγκόσμια πολιτική σήμερα. Το δεύτερο μέρος της ε, συνεδρίασης εστιάστηκε στο ζήτημα της οικονομικής διακυβέρνησης και στον καλύτερο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Εγώ ανέφερα το τι έχει κάνει μέχρι τώρα η ομάδα ε, στην οποία μου ζητήθηκε να προεδρεύσω. Ήδη υπάρχει μεγάλος βαθμός σύγκλησης και σκοπεύω η ομάδα αυτή να ολοκληρώσει το έργο της τον Οκτώβριο το αργότερο. Θα συναντηθώ με την αντιπροσωπεία σας και πριν και μετά τις διακοπές για να διασφαλίσουμε πως θα υπάρχει συνεισφορά του Κοινοβουλίου στο έργο μας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλωσόρισε την έκθεση προόδου την οποία έκανα και συμφώνησε σε κάποιους πρώτους προσανατολισμούς. Συμφώνησε πως θα πρέπει να υπάρχει αυστηρότερη επιτήρηση των προϋπολογισμών και της ανταγωνιστικότητας. Υπάρχει συμφωνία πως πρέπει να ενισχύσουμε και τις δύο πλευρές, και την προληπτική και την ε, διορθωτική πλευρά του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, οπότε προβλέπεται ένα σύστημα κυρώσεων για να έχουμε ένα συνεκτικό σύστημα. Επίσης συμφωνήσαμε στην ιδέα της Κομισιόν για ένα ευρωπαϊκό εξάμεινο, όπου τα κράτη-μέλη θα παρουσιάζουν ήδη την άνοιξη ε, προγράμματα σταθερότητας και σύγκλησης, για να μπορεί έτσι να γίνει μια κοινή αξιολόγηση των τάσεων των εθνικών προπολογισμών για τα επόμενα έτη, λαμβάνοντα βεβαίω βεβαίως υπόψη τι εθνικές διαδικασίες. Επ' αυτού, να τονίσω πως ποτέ δεν προτάθηκε οι Υπουργοί Οικονομικών να υποβάλουν τους προπολογισμού τους στην Κομισιόν προς έγκριση πριν πάνε στα Εθνικά Κοινοβούλια. Κανείς δεν θα τολμούσε μια τέτοια παραβίαση των κοινοβουλευτικών αρμοδιοτήτων το έργο της ομάδας μας αυτής δεν έχει τελειώσει. Άλλες ιδέες, από την Κομισιόν βεβαίω, από την Κεντρική Τράπεζα, από το Κοινοβούλιο σας και από τα κράτη-μέλη, από τα οποία είχαμε γύρω στις 12 γραπτές συνεισφορές, θα συζητηθούν ακόμα. Κάποιες από αυτές μπορούν να πετούν αλλαγή της συνθήκης. Αλλά επειδή αυτή είναι μια δύσκολη διαδικασία, θα δώσουμε προτεραιότητα στις προτάσεις εκείνες που μπορούν να πραγματοποιηθούν πιο γρήγορα και εύκολα. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται πως υπάρχει μια συνένεση για το ότι δεν χρειαζόμαστε νέα θεσμικά όργανα για την οικονομική διακυβέρνηση. Αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα αυτά τα οποία ήδη έχουμε. Και αν και ορισμένες φορές θα απαιτηθούν συγκεκριμένες αποφάσεις στο επίπεδο των χωρών της Ευρωζώνης, και όταν απαιτείται εγώ θα συγκαλέσω συνόδους της Ευρωζώνης όπως έκανα ήδη δύο φορές είναι στο επίπεδο του συνόλου της Ένωσης εκεί όπου πρέπει να αποφασιστούν τα της οικονομικής διακυβέρνησης. Είτε εντός είτε εκτός της Ευρωζώνης είμαστε οικονομικά αλληλένδετοι και από κοινού έχουμε τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου. Σε αυτό το επίπεδο πρέπει να λαμβάνονται οι περισσότερες ευρωπαϊκές ευρωπαϊκές αποφάσεις μέσω του θεσμικού πλαισίου της Ένωσής μας. Έτσι, σύμφωνα με την συνθήκη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σκοπεύει να εκπληρώσει τον ρόλο του, δηλαδή να δίνει πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες για την Ένωση και οικονομική στρατηγική. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη παραμένουν τεράστιες. Ήμασταν πολύ κοντά στο χείλος του γκρεμού πριν από λίγες εβδομάδες και ακόμα δεν είμαστε ασφαλείς. Δικαίως δώσαμε στο βαθύτερο σημείο της ύφεση οικονομική όθηση, αλλά πρέπει να προσέξουμε να μην φτάσουμε σημείο εκεί όπου τα ελλείμματα θα είναι πλέον αδύνατο να εξυπηρετηθούν και θα αρχίσουν να απειλούν την οικονομική μας ανάγκαψη. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν τα κρατη μέτρη για να μειώσουν τα ελλείμματά τους δεν θα έχουν αποπληθωριστικό αποτέλεσμα εάν αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία και άρα κινήσουν και την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Από την άλλη μεριά, εάν δεν διορθώσουμε μακροχρόνια ελλείμματα, θα οδηγηθούμε σε μοιραία απώλεια της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας κάτι το οποίο θα σημαίνει μακροπρόθεσμες οικονομικές ζημιές. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση του κάθε κράτους μέλους και είναι σταδιακά. Και μάλιστα αντί για το απόλυτο επίπεδο, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η κατεύθυνση και η βιωσιμότητα. Ή υπό την προπόθεση ότι θα επιμείνουμε, έχω την πεποίθηση πως η Ευρώπη θα στρίψει την γωνία, θα βγει από αυτή τη δύσκολη θέση. Θεωρώ λοιπόν πως αυτή η συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποτέλεσε άλλο ένα σημαντικό βήμα καταπολέμησης της κρίσης που ξεκίνησε ως χρηματοπιστωτική κρίση και έγινε οικονομική, δημοσιονομική και σχεδόν νομισματική κρίση. Αντλούμε λοιπόν τα μαθήματα τα οποία πρέπει και διορθώνουμε την πορεία μα βήμα προ βήμα. Είμαι πεπισμένο ότι θα επιτύχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το λόγο έχει ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, προεδρεύοντα, αγαπητά μέλη, συνάδελφοι, μία εβδομάδα πριν βρεθήκαμε στο Στρασβούργο για να προετοιμάσουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τη Σύνοδο των G20 στο Τορόντο. Τότε ανέφερα ότι η ανάπτυξη είναι η απάντηση στην οικονομική κρίση, η οποία θα πρέπει να μην είναι μια ευφυής απάντηση, θα πρέπει να βασίζεται στην φορολογική ολοκλήρωση. Και γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε σε διάφορα μέτωπα εισαγάγοντας τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 τακτοποιώντας τις εκκρεμότητες ως προς την χρηματοπιστωτική εποπτεία, ενισχύοντας την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη και μιλώντας ως Ευρωπαίοι με ενιαία φωνή στη Σύνοδο του Τορόντο των G20. Αυτή ήταν και η θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα με βάση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έφτασε σε ουσιώδη συμπεράσματα. Λάβαμε αποφάσεις για στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές που μας δίνουν ένα νέο όραμα τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν έχουν προσθετικό χαρακτήρα των εθνικών προοπτικών. Δίνουν μια ευρωπαϊκή προοπτική σε τρεις τομείς. Οικονομική διακυβέρνηση, ρύθμιση των χρηματοοικονομικών και εποπτεία και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 ως προς την οικονομική διακυβέρνηση έχει επιτελεστεί πρόοδος και έχουμε οριοθετήσει το θέμα. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Μαΐου υπέβαλε συγκεκριμένες ιδέες. Το Ευρωπαϊκό Εξάμειονο για, για τη σύγκληση των οικονομικών και φορολογικών πολιτικών πιο σωστή τακτική του καρότου και του μαστιγίου για αντιμετώπιση μελλοντικών προβλημάτων και διόρθωση αυτών και δημοσιονομικά πλαίσια που ορίζονται καλώς και συμβαδίζουν με τις συνθήκες καθώς και αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών στην εσωτερική αγορά για να καλύψουμε το πλήρες φάσμα των σημείων κλειδιών και να μην δούμε μόνο τη δημοσιονομική πτυχή. Τώρα υπάρχει μια ευρωπαϊκή συνένεση. Η Task Force και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να εμβαθύνουν αυτή τη συνένεση για να φτάσουμε σε λεπτομεριακές ε, δράσεις. Άρα την επόμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει ιδέες για συγκεκριμένη δράση και εργαζόμαστε επί των 10 προτάσεων που θα σας υποβάλουμε μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου γιατί έχει μεγάλη σημασία, έχει μεγάλη σημασία και τα χρονικά περιθώρια. Ο δεύτερος βασικός τομέας όπου επιτύχαμε συμφωνία, μια συμφωνία ήταν οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει η σωστή ρυθμιστική βάση έτσι ώστε να υπάρχουν υγιείς χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έτσι ώστε να μην υποκύψουμε στις μελλοντικές πιέσεις. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ιδιαίτερα σημαντικός όπως έκανα έκκληση και στους επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων, έτσι κάνω έκκληση και εσάς, έτσι ώστε να εγκριθούν οι χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές προτάσεις πριν από το καλοκαίρι, έτσι ώστε το σύστημα να τηθεί σε εφαρμογή πριν από το τέλος του επόμενου έτους, ως προς τις κεφαλουχικές ανάγκες. Χαίρομαι διότι θα αναλάβουμε τη νέα φάση των χρηματοπιστωτικών προτάσεων που θα εγκριθούν μέχρι το τέλος του 2011. Η Επιτροπή θα εστιάσει την προσοχή της προς αυτή την κατεύθυνση και το Κοινοβούλιο θα δώσει μεγάλη σημασία σε αυτή την σημαίνουσα πρωτοβουλία. Επίσης, είχε μεγάλη σημασία για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συμφωνήσει ως προς ε, ένα πραγματικό τεστ αντοχής για τις τράπεζες. Αυτό θα πρέπει να γίνει αναχρηματοπιστωτικό οργανισμό έτσι ώστε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και να ε, αποκόψουμε την κερδοσκοπία η οποία είναι ολέθρια για τις αγορές. Και όπως σας είπα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να γίνουν οι σωστές δοκιμές και παρεμβάσεις εκεί που κρίνεται αναγκαίο. Ένα άλλο βασικό σημείο της δράσης μας και ένα από τα βασικότερα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήταν η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, η οποία έγινε αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη όπως είχε προταθεί ορισμένους μήνες, λίγους μήνες πριν. Είμαι πεπισμένος ότι αυτή η προσέγγιση συμφωνήθηκε εντάχει διότι έτσι ακριβώς έπρεπε να γίνει, ιδιαίτερα ως προς τους πέντε στόχους για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση της εκπαίδευσης, διότι κάτι τέτοιο δεν ήταν σαφές εξ αρχής, ότι δηλαδή τα κράτη-μέλη θα ε, δεχτούν να ε, θέσουν σε ένα κοινό τραπέζι θέματα που είναι εθνικής αρμοδιότητας. Άρα οι 27 έφτασαν σε μακροχρόνιους στόχους και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχει μεγάλη σημασία η διακυβέρνηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα πρέπει να υπάρχουν αντιγνωμίες ως προς τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η μεγάλη όθηση που δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βοήθησε στην επίτευξη αυτού του θετικού αποτελέσματος και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ νέου, ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι κατά το πρώτο ε, τμήμα των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε το γεγονός ότι έπρεπε να επιτευχθεί συμφωνία επί των σημαντικών αυτών ε, θεμάτων. Σας ευχαριστώ για τη γενικότερη όθηση που δώσατε σε αυτούς τους στρατηγικούς στόχους, διότι όπως γνωρίζετε δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η εργασία. Θα πρέπει να ορίσουμε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα όπως την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής. Τώρα αντιμετωπίζουμε την, το θέμα της εφαρμογής της στρατηγικής. Θα πρέπει να συνταχθούν όλα τα μέρη της κοινωνίας γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να αναλάβουν αυτό το έργο και τα κράτη-μέλη. Δεν είναι μια στρατηγική που απορρέει από τις Βρυξέλλες ή το Στρασβούρο. Θα πρέπει να κινητοποιηθεί ολόκληρη η κοινωνία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβάλλει τις κατάλληλες στρατηγικές συνεργαζόμενοι από κοινού με τα κράτη-μέλη για να προβληθούν γενικότερες μεταρρυθμίσεις. Επίσης θα βασιστούμε στην εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ε, δικές σας εκλογικές περιφέρειες σε επίπεδο κοινωνικού ιστού και στην κοινωνία γενικότερα. Πρόκειται για κοινή προσπάθεια για τα για τους επόμενους μήνες και χρόνια. Έτσι έχουμε μία ευρύτερη, ευρεία, την ευρύτερη δυνατή πλατφόρμα για το Τορόντο, για τους G20, που μπορούμε να τους προσφέρουμε μετά το 2008 σε μία κοινή επιστολή του κυρίου Βαν Ρομπόη και εμού θα υποβάλουμε το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη συνάντηση. Είναι η πρώτη φορά που η Ευρώπη μιλά με μία φωνή σε σχέση με τις προτεραιότητές μας ως προς θέματα παγκόσμιας δράσης. Έχουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το μέλλον, δηλαδή οι προκλήσεις που θα προβάλλουμε και στους εταίρους μας Το θέμα δηλαδή του τραπεζικού φόρου και του φόρου τραπεζικών συναλλαγών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο φτάσαμε σε μια συνένεση σε αυτά τα ζητήματα. Εν συμπεράσματι μπορώ να πω ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δείχνει ότι είμαστε αποδετικοί όταν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με νέους μηχανισμούς και διαρθρώσεις τις προκλήσεις αυτές γιατί οι θεσμικές συζητήσεις δεν έχουν τέλους. Τέλος, θα πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς μας, γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε απτά αποτελέσματα, όπως κατέδειξαν οι εργασίες της ε, περασμένης εβδομάδας. Θα ήθελα να συγχαρώ το Κοινοβούλιο το Συμβούλιο και την ύπατη εκπρόσωπο για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Είναι αναπόσπαστο τμήμα των ευρωπαϊκών θεσμών μέσα σε μια συμφωνία της κάθε άστον και της Επιτροπής με βάση τους ίδιους κανόνες λογοδοσίας που ισχύουν για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση και εργαστήκαμε πολύ σκληρά έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να αρχίσει να λειτουργεί το ταχύτερο δυνατόν. Αυτή ήταν μία από τις βασικές καινοτομίες της συνθήκης της Λισαβόντς μπορείτε να βασιστείτε στην Επίτροπη για να φτάσουμε σε αυτά αποτελέσματα που αναμένουν οι πολίτες μας. Και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό αυτό το Συμβούλιο επιτέλεσε μεγάλες πρόοδους για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ομιλία σας και τώρα εκ μέρους των διαφόρων πολιτικών ομάδων θα ακούσουμε καταρχάς την κυρία Βόρτμαν Κόλ για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι Πρόεδροι, το ΕΛΚ είναι ικανοποιημένο για το το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπό την Προεδρία σας έκανε σημαντικά βήματα για την αναγκαία βελτίωση της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης και την κοινή στάση στους G20, αλλά η κρίση μας εξαναγκάζει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας πιο στέρεης βάσης για το ευρώ. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα μεγάλα προβλήματα για να αποκαταστήσουμε την αγορά των χρηματαγορών και των, και των ε, πολιτών μας. Εμείς στηρίζουμε την ενίσχυση του προληπτικού τμήματος ε, του Συμφώνου σταθερότητα και τι κυρώσει, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα προτείνει συγκεκριμένα η Task Force, γιατί η διακυβερνητική μέθοδος δεν θα μας βγάλει από την κρίση. Κατά την άποψή μας θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μια κοινοτική μέθοδο διακυβέρνησης. Κανένα νέο θεσμικό όργανο και σε αυτό συμφωνούμε, αλλά μια ανεξάρτητη και ισχυρή Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι καλό, κύριε Μπαρόσο, το ότι θα καταθέσετε τους ερχόμενους μήνες προτάσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα είπατε στο Κοινοβούλιο πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης και σας χειροκρότησε η Ολομέλεια. Πρέπει λοιπόν τώρα να φανείτε αντάξιος και φιλόδοξος του θεσμικού σας ρόλου. Ενίσχυση επίσης του δικαίου του ανταγωνισμού και στα 27 κρατημέλη. Αυτό θέλουμε να επιτύχουμε με τη στρατηγική του 2020, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως κινητήρα της ε, οικονομίας, αλλά και βεβαίως μετρώντας πώς θα συμπεριφερθούν τα κράτη-μέλη. Η δική μας η ομάδα σας ζητάει να καταλήξετε σε πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα επ' αυτού του σημείου στην Task Force. Αλλιώς κινδυνεύουμε να καταλήξουμε πάλι σε μια στρατηγική της Λισαβόνας η οποία δεν ήταν επιτυχημένη και αυτό δεν είναι προς το συμφέρον των πολιτών μας, των θέσεων εργασίας και της οικονομικής ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να αποφασίσετε σύντομα για το πακέτο οικονομικής επίβλεψης, αλλά ξέρετε πως το πρόβλημα δεν είναι εντός του Κοινοβουλίου. Το πρόβλημα είναι το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο δεν είναι διατεθειμένο να μετατρέψει την έκθεση Ντελαροζιέρ σε νομοθεσία. Δεν έχει υπάρξει αρκετή πρόοδος. Οπότε καλά θα κάνετε να παρακινήσετε και να απευθύνετε έκκληση στους συναδέλφους σας στο Συμβούλιο να είναι και αυτοί διατεθειμένοι για συμβασμούς όπως το Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να επιτύχουμε όπως είπατε τον στόχο του επομένου έτους. Τώρα η κυρία Ούλφ Σκοκ για τους σοσιαλιστές. Eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. 14.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως ε, χύνονται στον κόλπο του Μεξικού. Στη Βόρεια Ευρώπη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται ότι θα έρθει το πετρέλαιο και στις δικές μας ακτές. Είμαστε ιδιαίτερα ευάλωτοι σε τέτοιου είδους πετρελοκυλίδες. Και κανείς δεν ζει σε μια απομονωμένη νησίδα. Υπάρχει διασύνδεση. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να μην ξεχνούμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενέργειας και την ε, διαφοροποίηση Υπάρχουν πολύ καλά λόγια, πολλά ψηφίσματα που έχουν γραφεί, αλλά φαίνεται να μην γίνεται τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Και λόγω της οικονομικής κρίσης όλα αυτά τα αφήνουμε κατά μέρο, τα παραγνωρίζουμε. Αλλά δεν μπορούμε να επιλύσουμε την οικονομική κρίση αν δεν επιλύσουμε το ζήτημα της εξάρτησης, της ε, τροτότητας που έχουμε και της ε, ευάλωτης θέσης στην οποία βρισκόμαστε από ενεργειακής πλευράς τελικά βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν αυτοί είναι που πρέπει να πάρουν και τα μέτρα, να αντιδράσουν. Εδώ και δεκαετίες βλέπουμε ότι οι υπεύθυνοι διαφόρων πολιτικών ομάδων ήταν αυτοί οι οποίοι τελικά μιλούσαν ε, και προάσπιζαν ε, την ε, ανεξαρτησία και την κυριαρχία των χρηματοπιστωτικών αγών και τώρα λένε ότι πρέπει να ρυθμιστούν. Βλέπετε λοιπόν ποιε είναι οι συνέπειες της κατάστασης αυτής σε πολλά κράτη-μέλη, αυτού του άναρχου ανταγωνισμού και της πλήρους κυριαρχίας ε, των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών. Βλέπετε τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει αυτή η κατάσταση. Βλέπετε και τι δυσκολίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον μέχρι ότου αρχίσει να λειτουργήσει αυτός ο νέος μηχανισμός. Πώς θα μειωθούν τα ελλείμματα Κύριε Πρόεδρε, κινδυνεύουμε με παράλυση από όλη αυτή την κρίση. Κινδυνεύουμε να πέσουμε σε βαθιά ύφεση. Γι' αυτό λοιπόν σε όλα τα κράτη-μέλη είναι ανάγκη να δράσουμε έτσι ώστε να μην δημιουργήσουμε κοινωνικές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Να μην επιβαρύνουμε και επιδεινώσουμε ακόμη την κατάσταση που θέλουμε να σώσουμε. Άκουσα αυτά που είπε ο κύριος Φόνδρον Πάη και ο κύριος Μπαρόζα, αλλά τελικά ε, νομίζω ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν πιο πολύ με την αρχιτεκτονική, αλλά κυρίως θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα όχι μόνο τα οικονομικά αλλά και το περιβάλλον. Αν δούμε την ανεργία, την μαζική ανεργία η οποία αυξάνεται και σε αυτά τα μέτωπα πρέπει να δράσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, εκ μέρους των Φιλελευθέρων τώρα ο κύριος Φερχόφστατ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς επιτρέψατε μου να πω ότι είναι προφανές ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να διαδραματίσουν έναν σημαντικό, έναν ζωτικό θα έλεγα ρόλο στην οικονομική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης τα επόμενα χρόνια. Όμως υπάρχει και ένα άλλο σημαντικότερο ερώτημα. Το σημαντικότερο σήμερα ερώτημα είναι ποιος θα αναλάβει τον έλεγχο και ποιο θα επιβάλλει κυρώσεις εάν κάποιο από τα κράτη-μέλη δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις και τους όρους. Αυτό είναι το σημαντικό ερώτημα. Τον έλεγχο θα τον έχουν τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο. Θα αυτοκυρώνονται, θα αυτοτιμωρούνται τα κράτη-μέλη ή μήπως θα υπάρξει ένα κοινοτικό θεσμικό όργανο, ένα ανεξάρτητος θεσμός που θα αναλάβει τον έλεγχο. Αυτό είναι το σημαντικό ερώτημα σήμερα και πρέπει να σα πω ότι δεν νομίζω ότι εδώ στο Κοινοβούλιο υπάρχει έστω και ένα που να πιστεύει ότι τα κράτη-μέλη θα επιβάλλουν ε, κυρώσεις ε, στον εαυτό του. Μα δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα. Θα το κάνουν αγαπητοί συνάδελφοι στο μέλλον. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα. Γιατί απέτυχε η συνθήκη τη Λισαβόνα, Γιατί δεν υπήρχε σύστημα, δεν υπήρχε ένα ανεξάρτητο φορέα που να ελέγχει τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Το ίδιο γίνεται και με το σύμφωνο της ε, σταθερότητας και της ανάπτυξης. Όταν τα μικρότερα κράτη ε, δεν ε, εκπληρούσαν τις προϋποθέσεις, βιώναμε την ελληνική τραγωδία. Τι γινόταν όμως όταν μεγάλα κράτη σαν τη Γερμανία και τη Γαλλία, όταν αυτά οι μεγάλες χώρες δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, Εάν λοιπόν ε, θεωρήσουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, τότε θα πρέπει να το κάνει ένας ανεξάρτητος φορέας. Εμείς είμαστε πεπισμένοι για αυτό. Υπάρχουν μάλιστα και ψηφίσματα τα οποία εγκρίθηκαν σχεδόν ομόφωνα και πριν από δύο ημέρες νομίζω. Ο κύριος Τρισέο, Δεκαιτής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είπε ακριβώς αυτό. Έκανε ακριβώς την ίδια ανάλυση ενώπιον του Κοινοβουλίου αυτό το οποίο το Ευρωκοινοβούλιο, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, πιστεύει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Τρισέ μάλιστα πρότεινε έναν άλλο φορέα. Τέλος πάντων, εγώ δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε νέα θεσμικά όργανα, αλλά όπως και να έχει, βάσει της κοινοτική μεθόδου θα πρέπει ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο να ασκεί αυτόν τον έλεγχο. Όχι βέβαια ότι δεν θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν κάποιο ρόλο, θα πρέπει να υλοποιούν τη στρατηγική καθημερινώς ε, στο πλαίσιο των στρατηγικών που εκπονούνται σε επίπεδο κρατών μέλων. Αυτό χρειαζόμαστε λοιπόν. Χρειαζόμαστε ένα σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε στρατηγική 2020 και τη νέα στρατηγική που θα αναπτύξουμε για την ανταγωνιστικότητα. Και χρειαζόμαστε αυτόν τον έλεγχο. Δεύτερη παρατήρησή μου αφορά την ε, επίλεψη στον ε, χρηματοπιστωτικό τομέα. Βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για τη χρηματοπιστωτική επίβλεψη. Και ποιο είναι ο λόγο οι Υπουργοί Οικονομικών του ΕΚΟΦΗΝ το Δεκέμβριο ουσιαστικά δεν υιοθέτησαν την έκθεση Λαροζιά και τι προτάσεις της Κομισιόν. Εκείνη το πρόβλημα. Θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στους Υπουργούς Οικονομικών. Πρέπει να μελετήσουν εκ νέου τις προτάσεις τους, να επαναχωρήσουν και να ακολουθήσουν ε, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή για τις Τράπεζες. Αυτή ουσιαστικά είναι η πρόταση. Και αυτό το οποίο έκαναν οι Υπουργοί Οικονομικών στο ΕΚΟΦΗΝ του προηγούμενου Δεκεμβρίου ουσιαστικά ήταν ένα είδος συντονισμού κάποιο συντονισμό. Μα αυτό δεν έχει λειτουργήσει, δεν απέδωσε στην χρηματοπιστωτική αυτή κρίση. Κανένας δεν έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου. Τώρα λέμε ότι είναι καλό το σύστημα και ότι απλά χρειάζεται συντονισμό. Όχι βέβαια. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν από το Συμβούλιο, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπάρχει πίεση. Αυτό πρέπει να γίνει. Να ασκηθούν πιέσει στα κράτη-μέλη για να κινηθούν προ την κατεύθυνση μια ευρωπαϊκή εποπτική αρχή βάσει των προτάσεων τη έκθεση Λαροζιέρα. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. President. On behalf of, uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους των Πρασίνων ε, και της Ελεύθερης Μαχίας η κυρία Ρεμπέκα Χάρμ, συμπρόεδρος. Ähm, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, πρώτα απ' όλα να πω πως εξεπλάγει που είπατε πόσο φυσιολογική ήταν η σύνοδος προηγούμενης εβδομάδας είναι η συνέχεια της λανθασμένης μεθόδου της προηγούμενης εβδομάδας. Δεν θα πρέπει να παριστάνουμε πως έχουμε φτάσει σε φυσιολογική κατάσταση στην ευρωπαϊκή συνεργασία όταν περιορίζεται μία σύνοδο σε έξι ώρες για να μην πει κανείς καμιά λάθος λέξη και καταρρεύσει το ευρώ. Αυτό κυκλοφορούσε στο κτίριο του Συμβουλίου και δεν πρέπει νομίζω να είναι η δική σας η δουλειά να μας ρίχνετε στάχτη στα μάτια. Νομίζω μπορούμε να δούμε καθαρά τα πράγματα. Κυρίε και κύριοι, ο κύριος Φερχόφστατ είπε ήδη πως δεν πάνε καλά τα πράγματα με την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση και πως μπορούμε σε συγκεκριμένα πράγματα ήδη να το δούμε αυτό. Να το τονίσω. Οικονομική επιτήρηση και η έκθεση Λαροζιέρα αναφέρθηκαν. Κύριε Μπαρόζο, κύριε Φανρόμποη, τι άποψη έχετε για το ότι μετά από ένα χρόνο συζήτηση συμφωνήσαμε τώρα για την εποπτεία, αλλά το Συμβούλιο αρνείται να δώσει σε αυτή την εποπτεία δυνατότητες παρέμβασης. Και αυτό είναι μόνο στο επίπεδο των κρατών μελών. Αυτό είναι παράλογο. Ειδικά όταν σας στηρίζουμε εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περιμένουμε περισσότερα. Μπορούμε να συζητήσουμε τη συζήτηση για το τι θα ήθελε να επιτύχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απαγόρευση επικίνδυνων προϊόντων που υπάρχουν στις χρηματαγορές. Τουλάχιστον για την προσωρινή τους απαγόρευση. Μπορούμε να συζητήσουμε επίσης για το τι γίνεται με τα hedge funds και τους φορολογικούς παραδείσους για τους μισθούς των μάνατζερ και τα τεράστια μπόνους που πληρώνονται εκεί πέρα. Σε όλους τους τομείς γίνεται τριμερής διάλογος και παντού μπλοκάρει είτε το Συμβούλιο ή Συμβούλιο και Κομισιόν μαζί τα πράγματα. Και κύριε Μπαρόζο, μας ευχαριστήσατε για το ότι εμείς ως Κοινοβούλιο σας υποστηρίξαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Σωστό είναι αυτό η προσέγγιση αυτή του Κοινοβουλίου για την κοινοτική μέθοδο. Αλλά εάν δούμε πάλι τι γίνεται με το φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ε, θα ήθελα να ελπίζω πως κάτι θα γίνει στους G20. Αναμένω να έρθετε από το Τορόντο. Εάν επιστρέψετε και έχετε κάτι να μας φέρετε, φροντίστε τουλάχιστον ο αρμόδιος επίτροπος να έχει την ενιαία ευρωπαϊκή θέση. Το λέει και ο κύριος Γιούνκερ συνέχεια. Επιτέλους να υποβάλει κανονική πρόταση για την εισαγωγή του αυτού του φόρου στην Ευρωζώνη. Και εάν όχι, τότε σπαταλήσατε άλλη μία σύνοδο για να δείξετε στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη τι, ότι υπάρχει και αυτό το μέσο. Τώρα για τη στρατηγική της ε, Ευρώπης 2020, αν δούμε την Ελλάδα ή την Ισπανία, πρέπει να υπάρχει μια κοινή στρατηγική που θα δώσει τον προσανατολισμό για το πώς θα επιτύχουμε την βιώσιμη ανάπτυξη. Καλό θα ήταν να υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά τι έχουμε εμείς εδώ πέρα. Έχουμε ωραία λόγια, ωραιότερα από τη στρατηγική της Λισαβόνας, αλλά για τα ωραιότερα αυτά λόγια, η φόρο ανάπτυξη, ε, το ακούμε συνέχεια πια εδώ μέσα, ε, μας λείπουν όπως και από τη στρατηγική της Λισαβόνας τα μέσα και τα λεφτά. Και αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση σε μένα ως πράσινη, δεν υπάρχει πεποίθηση για το ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε ενεργειακή αποτελεσματικότητα, αποτελεσματική χρήση πόρων, σοβαρή προστασία του κλίματος και για το ότι όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν κινητήρα της καινοτομία. Αυτή τη στιγμή στη Γερμανία πανηγυρίζουν για το ότι ανακάμπτει η αυτοκίνητο αυτοκινητοβιομηχανία γιατί οι Κινέζοι αγοράζουν μεγάλα αυτοκίνητα με πολλούς ύπους που καίνε πολύ βενζίνη. Αυτό αφού έγινε η καταστροφή με το πετρέλαιο και της προαναγγελθήσας αποτυχίας του Κανκούν. Νομίζω δεν έχουμε καταλάβει καν στην Ευρώπη τι εστί βιώσιμη ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ Κέρκοπ για τους συντηρητικούς. Κύριοι Πρόεδροι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δικαίως επικεντρώθηκε στη μεταρρύθμιση της Ευρώπης, κάτι το οποίο υποστηρίζει και η ομάδα μου. Αλλά θα ήθελα πρώτα να πω κάτι για το Ιράν. Το Ιράν, κύριε Πρόεδρε, θα έπρεπε να είναι μία από τι πιο σεβαστέ δυνάμει στη Μέση Ανατολή. Έχει μία μακρόχρονη ιστορία και ένα λαό ο οποίο είναι καινοτόμο και ταλαντούχος. Και θα θέλαμε να συνεργαστούμε με το Ιράν, το Ιράν για να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα παγκόσμια προβλήματα. Συναντήθηκα πρόσφατα με εκπροσώπους του Ιράν που πρότειναν μερικά από αυτά τα ζητήματα. Αλλά δυστυχώ, κύριε Πρόεδρε, το Ιράν είναι στα χέρια εκείνων που δεν ενδιαφέρονται για τι φιλοδοξίε του ίδιου τους του λαού ή τι ανησυχίε των γειτόνων στον κόλπο. Χωρί περίσκεψη ακολουθεί ένα πρόγραμμα πυρηνική ενέργεια που δικαίω γεννά υποψίε. Εάν ανέπτυσε την πυρηνική ενέργεια με τρόπο διαφανή, κανεί δεν θα αμφισβητούσε το δικαίωμά του να το κάνει. Αλλά με το να προσπαθεί να απτύξει αυτέ τι δυνατότητε έγκρυπτο, δεν υπάρχει αμφιβολία πως τα κίνητρα και οι φιλοδοξίες του είναι επικίνδυνες. Οπότε καλωσορίζουμε τα βήματα τα οποία έλαβαν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αυξήσουν την πίεση και να συνεργαστούν με την παγκόσμια κοινότητα. Εάν δεν γίνουν αυτά, δυστυχώ θα πρέπει να ληφθούν μέτρα στον τομέα των μεταφορών της ε, βιομηχανίας του αερίου και του τραπεζικού τομέα. Επίση, καλωσορίζουμε τη στρατηγική του 2020 που δικαίω θεωρείται το κύριο έργο τη Κομισιόν. Δεν συμφωνούμε με κάθε λεπτομέρεια, αλλά εάν τα λόγια γίνουν πράξη θα έχουμε θετική εξέλιξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αποκατασταθεί και θα επεκταθεί η ενιαία αγορά. Πρέπει επίσης να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί το εμπόριο εντός και εκτός, να απομακρυνθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, να μειωθούν τα βάρη στις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες. Η δε ρύθμιση πρέπει να αντικατασταθεί και από βαριά, να γίνει έξυπνη ή και λιγότερη. Για χάρη του ευρώ και του οικονομικού μέλλοντος όλων των χωρών Τη Ένωση. τα ε, ελλείμματα του υπερβολισμού πρέπει να μειωθούν βεβαίω σε όλε τις χώρες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και εμεί με τη σειρά μα λαμβάνουμε αυτά τα επώδυνα αλλά αναγκαία μέτρα. Ο προπολογισμό, εκτάκτου ανάγκη, όπω ανακοινώθηκε χθε ήταν δραματικό, αλλά όπω είπε ο Υπουργό Οικονομικών αναπόφευκτος. Μόνο μειώνοντα το δημόσιο χρέο και έχοντα χαμηλά μακροπρόθεσμα επιτόκια θα μπορέσει ο, δημόσιος, ο ιδιωτικό τομέα να επενδύσει και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Και ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να μας οδηγήσει στην ανάπτυξη και την ευημερία. Καλωσορίζουμε το ότι το Συμβούλιο έλαβε άμεσα πρακτικά βήματα για να στηρίξει το ευρώ. Βεβαίως η χώρα μου δεν είναι στο ευρώ και δεν θα μπει, αλλά θέλουμε να είναι επιτυχημένο το ευρώ. Αλλά η ομάδα μας πιστεύει πως τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για τη διακυβέρνηση του ευρώ δεν απαιτούν περισσότερη κεντρική διοίκηση και εμείς δεν θα θέλαμε να οδηγηθούμε σε μεταβίβαση εξουσιών από τα κράτη-μέλη στι Βρυξέλλε. Ούτε να υποχρεωθούν κράτη που δεν είναι μέλη του ευρώ να στηρίξουν την Ευρωζώνη. Κάτι το οποίο είναι κυρίω ευθύνη των κρατών μελών τη Ευρωζώνη. Βεβαίω υποστηρίζουμε πρωτοβουλίε που σέβονται τι συμβατικέ υποχρεώσει των κρατών μελών μα. Κύριε Πρόεδρε, ζούμε σε μια ανταγωνιστική εποχή. Η περίοδο τη οικονομική κυριαρχία τη Ένωση και των ΗΠΑ προφανώ τελειώνει το σύστημά μας της ελεύθερης αγοράς, φιλελεύθερης δημοκρατίας φαίνεται πως κινδυνεύει από άλλους που την προς ένα πιο αυταρχικό καπιταλισμό. Γι' αυτό θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε για να μπορούμε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τον ελεύθερο τρόπο ζωής μας. Το να προσπαθούμε να αποδράσουμε από αυτή την ανάγκη με το να επιμείνουμε στο status θα ε, μας οδηγήσει οπωσδήποτε στην καταστροφή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα αποτελέσματα του Συμβουλίου της Πέμπτης πρέπει να μετρηθούν σε σχέση με τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προκλήσεις. Είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις αιτίες της ε, κρίσης που ξεκίνησε από τις ε, αρχές Μαΐου. Ποιες προτάσεις ε, κάνετε στους Ευρωπαίους πολίτες και στις χρηματαγορές για να αποκατασταθεί η λειτουργία του συστήματος. Το Συμβούλιο λέει πως αυτοί προκάλεσαν την κρίση οι τράπεζες, δηλαδή να συμμετάσχουν, να πληρώσουν και να ρυθμιστούν οι δραστηριότητες τους. Αυτό το χαιρετίζω αλλά δεν το πιστεύω γιατί αποφασίζουν πρώτα απ' όλα μια διεθνή τραπεζική εισφορά για την οποία ούτε καν με στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει συμφωνία και την οποία πέριψαν τελείως κάποιες χώρες του G20. Οπότε το να περάσει αυτή η απόφαση δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό. Δεύτερον, για την εισαγωγή γενικού φόρου ε, στις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές υπάρχει μια διερευνητική εντολή. Δεν ξέρω εάν μπορούν έτσι να καθυσυχαστούν οι αγορές ή να σταματήσει η κερδοσκοπία ή βεβαίω εάν μπορεί να ληφθεί μια τέτοια απόφαση στους G20. Τρίτον, τα αυστηρότερα μέτρα κατά των ελλημάτων σε μια χρηματοπιστωτική κρίση μάλλον θα χειροτερεύσουν τα πράγματα, θα μειωθεί η κατανάλωση των πολιτών και ιδιαίτερα θα πλήξουν τους οικονομικά ασθενέστερους οι οποίοι θα σφίξουν περισσότερο τη ζώνη. Οπότε έχει προγραμματιστεί η συνέχεια από εδώ και μπρος. Θα απαιτηθούν και νέα μέτρα εξοικονόμησης, κάτι το οποίο θα αμφισβητήσει πλήρως στρατηγική για την Ευρώπη 2020 και τέλος θα συρρυκνωθεί η πηγή εσόδων των ε, κρατών μελών. Ενώ θα έπρεπε αυτή να ενισχυθεί μέσω ευρωομολόγων ή κοφόρων, όλα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη. Κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο. Πέμπτον, η κρίση αυτή υποσκάπτει τη δημοκρατική βάση της κοινωνίας μας. Και βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα μειώσεις ε, του κοινωνικού κράτους, μισθών και συντάξεων, αύξηση των ε, ορίων συνταξιοδότησης και το αποτέλεσμα είναι ότι ανοίγει συνεχώς η κοινωνική ψαλίδα και πλήττονται μόνο οι φτωχοί. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα από την ε, Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας ο κύριος Φαν Ράμπα, ο κύριος Κύριε Φαν Ράμπα, σας ευχαριστούμε πολύ για την ε, ομιλία σας. Είπατε ότι έγινε η διάσκεψη κορυφής, ότι έφυγε η οικονομική κρίση, ότι φύγαμε από το χείλος της καταστροφής και μετά μας δώσατε το σλόγγαν της ημέρας λέγοντας ότι το ευρώ ήταν θύμα της επιτυχίας του. Τουλάχιστον αυτό θα κάνει να χαμογελάσουν ε, πολλοί ε, πολίτες της Ευρώπης όταν δουν ή ακούσουν τις ε, είστε πραγματικά ένας όνειρομπόλος. Ε, σας προειδοποίησαμε από την αρχή ότι πολλές χώρες δεν μπορούν στην Ευρωζώνη. Δυστυχώς το ξέρατε, ξέρετε ότι εξαπάτησαν, ότι είπαν ψέματα, αλλά παρόλα αυτά ε, μπήκαν στην Ευρωζώνη. Σαν τον Ίκαρο, ο οποίος με τα κέρινα φτερά και ξέροντας ότι θα αλλιώσουν στον ήλιο, ανέβαινε ψηλά με τα φτερά. Και έπεσε βέβαια. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο άλλο σχέδιο, κάποιο εναλλακτικό σχέδιο για χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία που σε κάποια στιγμή θα χρειαστεί να εγκαταλείψουν το κοινό νόμισμα. Δεν υπάρχει άλλο σχέδιο για να επανέλθουν στο παλαιό εθνικό νόμισμά τους. Πόσο θα πρέπει να υποφέρουν αυτές οι χώρες ε, κυνηγώντα το ευρωπαϊκό όνειρο τι επίπεδο ε, κοινωνικών, ταραχών είναι αποδεκτό για να διατηρηθεί ένα κοινό νόμισμα που δεν αποδίδει, δεν έχει αποτέλεσμα. Διερωτώ με πόσο θα συνεχίσουν να πληρώνουν του τεράστιου λογαριασμού οι Γερμανοί. Αυτό που είναι τρομερό είναι ότι όλοι εδώ στην αίθουσα ε, πιστεύουν ότι το κάνουμε όλο αυτό για να είμαστε καλοί Ευρωπαίοι. Εγώ θα σας το πω. Καμία σχέση με την Ευρώπη δεν έχει αυτό το μέρος. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ταυτότητα η ισχύ της Ευρώπη ουσιαστικά έγκυται στην πολυμορφία της, στι γλώσσε της, στου πολιτισμούς της και στα κράτη της. Και ε, η ειρωνία είναι ότι εμείς οι ευρωσκεπτικιστέ είναι αυτοί οι οποίοι θα καταλήξουμε να είμαστε καλοί Ευρωπαίοι. Σα ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριο ε, Μαντλένερ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω πως είμαι ικανοποιημένος για το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ολλανδία γιατί το κόμμα μου πήγε από τις 9 στις 24 έδρες το κόμμα για την ελευθερία. Γιατί, γιατί οι Ολλανδοί θέλουν λιγότερη μετανάστευση, περισσότερη ασφάλεια και λιγότερη Ευρώπη πάνω απ' όλα. Η εσωτερική αγορά λειτουργεί μια χαρά, αλλά η μεταβίβαση χρημάτων από τα πλούσια ασθενέστερα κράτη πρέπει να σταματήσει. Και εδώ πέρα κύριε Φανεροπαϊσούλτς και Μπαρόσο τα πράγματα πάνε στραβά. Την δε επέμβαση αυτή έπρεπε να την είχατε κάνει εδώ και χρόνια όταν μπήκε η Ελλάδα με ψεύτικα νούμερα. Ήσασταν τυφλοί, τυφλοί γιατί θέλατε μόνο να επεκταθείτε και εξακολουθείτε να είστε. Και βλέπετε τώρα τι χώρε χτυπάνε την πόρτα μα. Η Αλβανία, το Κόσοβο, Βοσνία, Τουρκία. Και σήμερα μιλάτε και για την Ισλανδία. Μια χώρα χρεοκοπημένη. Η οποία από ό,τι φαίνεται είναι και υπέρ της αλληλείας φαλενών. και από ό,τι φαίνεται οδήγησε και ευρωπαϊκές τράπεζες στο χείλος του γκρεμού. Και εσείς λέτε στην Ισλανδία ελάτε και να συνεχίσετε και τι απάτε και να συνεχίσετε να σκοτώνετε κεφάλαιε. Έχετε τυφλωθεί από την επιθυμία σας για διεύρυνση και δεν εξυπηρετείτε τις πολίτε μας. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Άκουσα έναν βουλευτή να λέει ότι αυτό το κοινοβούλιο δεν είναι ένα πραγματικό κοινοβούλιο αλλά ένα ψεύδο κοινοβούλιο. Άρα τι δουλειά έχει εδώ και πόσοι φορολογούμενοι πληρώνουν το δικό του μισθό. Κύριε Πρόεδρε, να είμαι ξεκάθαρος. Τι κάνουμε εδώ πέρα. Αντιπαλεύουμε ανθρώπους σαν και εσάς και υπερασπίσουμε τι ευρωπαϊκέ αξίε έναντι ενό κοινοβουλίου που σπαταλά χρήματα. Και το αποδείξαμε, ο λαό μα εμπιστεύτηκε, κερδίσαμε σε εκλογέ και τι επόμενε φορέ θα έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Λοιπόν, θα δώσω τώρα το λόγο στον ε, κύριο Χέρμαν Φον Ρόμπαϊ, τον πρόεδρο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, δεν ε, έχω πρόβλημα μεγάλο τουλάχιστον με διάφορες επικρίσεις, αλλά με τη γενική προσέγγιση έχω πρόβλημα και εξηγούμε. Όταν ήρθα εδώ το Φεβρουάριο ή αρχές Μαρτίου, όταν μιλούσαμε για τα αποτελέσματα του πρώτου άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπήρχαν έντονες αμφιβολίες ότι θα επιτύχουμε να δημιουργήσουμε για την Ελλάδα ένα σχέδιο οικονομικής στήριξης και ότι η Ελλάδα θα είναι σε θέση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσει τα κακά του παρελθόντος. Υπήρχαν έντονες αμφιβολίες και κάποιες εβδομάδες μετά υπήρχε αυτό το σχέδιο το 110 δις ευρώ και είχε η Ελλάδα κάνει μεγάλη προσπάθεια τουλάχιστον για 10% του ΑΕΠ για να διορθώσει τα πράγματα, τα δημοσιονομικά της και κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να τα καταφέρει. Όταν πριν από κάποιες εβδομάδες είχαμε πει ότι θα δημιουργήσουμε ένα σχέδιο διάσωσης δυνητικής ύψος 750 δις, ε, των οποίων τα 500 προέρχονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη, δεν θα μας πίστευαν. Αλλά έγινε παρόλα αυτά. Είπαν κάποιοι. Μα οι χώρες της Μεσογείου έχουν ε, μια άλλη κουλτούρα. Δεν είναι σε θέση να πάρουν πραγματικά μέτρα μεταρρύθμιστης. Είναι χαμένος χρόνος και κόπος. Όταν βλέπω όμως αυτό που γίνεται σήμερα στις χώρες αυτές ε, και σε πραγματικά επώδυνες συνθήκες, Φυσικά και δεν χαίρεται κανείς γι' αυτό, αλλά βλέποντας αυτά που γίνονται σήμερα, εγώ πραγματικά βλέπω ότι υπάρχει μια βαθιά αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας. Όταν ακούω κριτικές και επικρίσεις για το κλίμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα στον κόσμο. Και δώσαμε μάλιστα σε αυτό το πρόγραμμα 20-20-20 και την απαραίτητη στήριξη και χρηματοδότηση και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι και τη νομική βάση. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν κάνουμε τίποτα. Φυσικά και δεν πρέπει να υποπέσουμε στο αμάρτημα της αυταρέσκειας σε καμία περίπτωση. Θεωρώ όμως ότι Κάποιοι θεωρούν ότι οτιδήποτε καταφέρνουμε είναι πολύ λίγο, πολύ αργά και ουσιαστικά ασήμαντη ε, επιτυχία. Όχι, πρέπει να αναγνωρίσουμε τα θετικά αποτελέσματα που είχαν οι δράσεις μας. Όταν ε, μιλάμε για καλύτερη διακυβέρνηση. Φυσικά. Φυσικά. Το ευρώ μας βοήθησε τα μάλα στη χρηματοοικονομική κρίση. Ούτε για ένα δευτερόλεπτο δεν θέλω να φανταστώ ποιε θα ήταν οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης αν δεν είχαμε στη διάθεσή μας αυτό το κοινό νόμισμα για 350 εκατομμύρια. Δεν μπορώ να φανταστώ καν τι θα γινόταν από πλευράς νομισματικής αστάθειας αν δεν υπήρχε το ευρώ. Θα είχαμε γυρίσει στην κρίση της δεκαετίας του 30 με την ε, υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και με τις καταστροφικές πολιτικές beggar my neighbor ο, γείτονα, ο, Σιτιάνος γειτονάς μου. Υπάρχουν βέβαια σίγουρα και αποκλήσεις και διαφορές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Δεν ήμουν εδώ ε, τις 10, τα δέκα πρώτα χρόνια του αιώνα μας, κάπου αλλού ήμουνα, αλλά ποιος εδώ, στο ημικύκλιο ή εκτός σε κάθε είδους ε, θεσμικό όργανο ή άλλο φορέα. Ποιος επισήμανε τόσο σημαντικά προβλήματα ε, ισοζυγίου πληρωμών ανταγωνιστικότητας. Λίγοι κανένας. Τώρα όμως ε, δικάζουμε για λάθη του παρελθόντος. Κοιτάξτε, είναι συλλογική η αλλο φορεα ποιος επισημανε τοσο σημαντικα προβληματα ισως υγιου πληρωμων ανταγωνιστικοτητας λιγοι κανενας τωρα ομως δικαζουμε για λαθη του παρελθοντος κοιταξτε ειναι συλλογικη η ευθυνη που έχουμε. Επομένως, για να είναι το ευρώ ένα σταθερό νόμισμα θα πρέπει η οικονομική και πολιτική ανάπτυξη, η οικονομική και η κοινωνική πολιτική να συγκλίνουν περισσότερο. Και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και σε ό,τι αφορά την πολιτική και ακριβώς αυτό το έργο προσπαθούμε να επιτελέσουμε. Κυρώσεις. Εγώ επιμένω να πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά άλλα επιχειρήματα αντί των κυρώσεων που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Οι κυβερνήσεις δεν δρούν με πρώτο κριτήριο το φόβο της κύρωσης στην Task Force θα εργαστούμε και θα προσπαθήσουμε να συγκεκριμενοποιήσουμε τις κυρώσεις όχι μόνο για διορθωτικές κινήσεις, δηλαδή για όσους υπερβαίνουν το 3% σε ό,τι αφορά το έλλειμμα, αλλά και για προληπτικούς λόγους, για όσους είναι κάτω από το κατόφλι αυτό του 3%, αλλά δεν σέβονται το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμά τους και των οποίων ε, το χρέος είναι ιδιαίτερος υψηλό και δεν φαίνεται να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση ή δεν γίνονται επαρκείς προσπάθειες. Θα εισαγάγουμε λοιπόν στο βαθμό που μας το επιτρέπει η συνθήκη κυρώσει οι οποίες υπερβαίνουν το σχέδιο και το σύμφωνο σταθερός και ανάπτυξη που έχουμε τώρα θα θεσπίσουμε αυτές τις κυρώσεις ε, στο ε, προληπτικό κομμάτι και θα τις ενισχύσουμε στο διορθωτικό κομμάτι. Δεν θα εφεύρουμε κυρώσεις που δεν έχουν καμία νομική βάση μέσα στη συνθήκη. Δεν ε, γίνεται αυτό, ούτε καν θα το σκεφτώ. Και αγαπητοί συνάδελφοι, για πρώτη φορά, γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα, θα θεσπίσουμε μηχανισμούς για την έλλειψη ισορροπίας, για το ισοζύγιο πληρωμών, για άλλα θέματα και για την μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Για πρώτη φορά θα γίνει κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν το είχαμε επιχειρήσει μέχρι τώρα. Θα καινοτομήσουμε λοιπόν με αυτήν την task force και αυτό χάρη στις ιδέες και στις προτάσεις και στις πρωτοβουλίες που θα μας κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προσεχείς εβδομάδες στον κρίσιμο αυτό τομέα της ανταγωνιστικότητας. Επομένως πραγματικά, πραγματικά αντιτίθεμε, αντιτίθεμε σε αυτόν ε, τον ε, ευρωσκεπτικισμό ο οποίος θέλει να ανατρέπει τα πάντα ενώ υπάρχουν προγράμματα υπάρχουν προθέσεις να μας ε, κατηγορούν και να μας ε, απορρίπτουν ε, εκ των προτέρων. Κάνουμε μεγάλη πρόοδο, κάνουμε βήματα στον τομέα της διακυβέρνησης, βήμα-βήμα, σταδιακά, αλλά είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, χρηματοπιστωτική εποπτεία, φυσικά, φυσικά και το συζητούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Φυσικά και το συζητούμε και με τους Υπουργούς Οικονομικών. Αλλά ξέρετε εδώ τώρα είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορούμε να μιλήσουμε για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία και εδώ δεν είναι αμαρτία, ούτε γίνεται κακό προαίρετα. Δεν θέλουμε να κάνουμε κηρύγματα, ούτε να δώσουμε μαθήματα σε κανέναν. Απλά συζητούμε και ούτε θέλω να διακομωδήσω ή να γελιοποιήσω τις προτάσεις που γίνονται και ότι θα τις πετάξουμε στα σκουπίδια. Όχι, εγώ δεν κάνω τέτοιου είδους ε, διακομωδήσεις και γελιοποίησεις. Κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλα ε, ζητήματα στο γραμματοψηφιακό τομέα, αλλά σε αυτό το πολύ κρίσιμο τομέα πρέπει να συνεργαστούμε, πρέπει να εργαστούμε μαζί. Συμβούλιο, ούτε καν Συμβούλιο Ευρωπαϊκό, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε την πρώτη η καταληκτική ημερομηνία, να μπορέσουν να ξεκινήσουν ε, αυτοί οι νέοι φορείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, στο χρηματοπιστωτικό τομέα. εδώ η Ευρώπη έχει τα ενία. Είναι, θα έλεγα, σκαπανέας. Αν όλες οι νεοι φορεί. αυτο ειναι παρα πολυ σημαντικο τωρα στο χρηματοπιστωτικο τομεα και εδω η ευρωπη εχει τα ενια ειναι θα ελεγα σκαπανεα αν όλε οι συμμετέχουσε χώρε. οι χωρες που συμμετέχουν ε, στην ε, G20, τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πρόεδρος Μπαρόζο και εγώ, αν προτείνουμε ένα τραπεζικό φόρο, τι θα γίνει, πιστεύετε ότι θα μας χειροκροτήσουν. Είμαστε όμως καπανείς, είμαστε καινοτόμοι και σε αυτό τον τομέα. Εμείς δείχνουμε τον τρόπο, τον και τον δρόμο. Θα είμαστε και για το φόρο για τις χρηματοπιστωτικές αλλαγές οι πρόδρομοι, οι σκαπανείς. Επομένως και σε αυτούς τους τομείς λαμβάνουμε στεναρές, θαραλές πρωτοβουλίες και θα τις προασπίσουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και σε κάποιους τομείς, όπως είναι ο τραπεζικός φόρος, το έχουμε πει και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν δεν υπάρξει συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο, θα δραστηριοποιούμε, θα δράσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη κάποια κράτη-μέλη λαμβάνουν πρωτοβουλίες, εγώ είμαι υπερήφανος και ευτυχής. Ήμουν κατά τον παρελθόν ε, και εμείς νομίζω είμαστε οι μόνη ίσω ή τέλο πάντων η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που λάβαμε τη σχετική πρωτοβουλία για έναν φόρο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Άκουσα πολύ καλά. Έλαβα υπόψη μου τα όσα άκουσα, αλλά θεωρώ ότι μια καλή προσέγγιση είναι μια θετική προσέγγιση. Ορισμένοι από εσά μα παροτρύνουν να είμαστε πιο θετικοί, ενώ συγχρόνω μα επικρίνεται. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Θα ήθελα ωστόσο σε κάθε περίπτωση να τονίσω αυτό το οποίο καταφέραμε, αυτό που πετύχαμε μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες αυτά, αυτούς τους τρεις-τέσσερις πρώτους μήνες της χρονιάς. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Και είμαι πεπισμένος ότι μετά από κάποιους μήνες αυτοί οι οποίοι είναι επικριτικοί σήμερα θα μας δικαιώσουν αν δεν μας χειροκροτήσουν. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Παρόζο. Ευχαριστώ. Σε σχέση με το ειδικό ερώτημα που μου ετέθη ως προς το πακέτο χρηματοπιστωτικής εποπτείας, αυτή η χρηματοπιστωτική εποπτεία είναι αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής μεταρρύθμισης, διότι οι νέες αυτές διευθετήσεις αφορούν το νέο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Προτείναμε η οίκη αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να την χάνουν ελέγχου, κάποιο ελέγχου από έναν φορέα. Γι' αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουμε ως προς αυτό το εποπτικό οικοδόμημα που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζήτησε από την Επιτροπή Ψηλού Επιπέδου υπό την ηγεσία του, του κυρίου Ντελαροζιέρ να μου υποβάλει τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε το Συμβούλιο να αλλάξει από την αρχική θέση του Δεκεμβρίου ως προσορισμένα βασικά σημεία, τα οποία θεωρήσαμε πολύ σημαντικά και εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να επιτύχουμε έναν συμβιβασμό. Εδώ θα πρέπει να ασκηθεί πίεση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν παραμείνουμε σε μία θέση όπου θεωρούμε ότι ο γείτονα δεν κάνει αρκετά, τότε δεν θα προχωρήσουμε. Πρέπει να επιτύχουμε ένα συμβιβασμό. Και πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μία συμφωνία ακολουθώντας και συμπορευόμενοι με τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να υπάρξει μία, ένας φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών Επίσης, να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα προς τις επιχειρήσεις, προς τη στήριξη επιχειρήσεων μέσα στα πλαίσια αυτών των συναλλαγών και ένα ταμείο εγκυοδοσίας καταθέσεων. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Αύριο θα προωθηθεί ένας τριμερής διάλογος που έχει μεγάλη σημασία. Εάν καθυστερήσουμε τα πράγματα δεν θα γίνουν πιο εύκολα. Γιατί πολλοί που εκφράζουν επιφυλάξεις θα προβάλλουν δυσχέρειες. Νομίζω όμως ότι τη στιγμή που θέλουμε ένα ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν πρέπει να αναβάλουμε κάτι τέτοιο, διότι μία πλήρης δεύτερη ανάγνωση δεν θα μας επιτρέψει να αρχίσουν να λειτουργούν αυτοί οι φορείς από την 1η Ιανουαρίου 2011. Γι' αυτό και υπάρχει επίγον χαρακτήρας να έχουμε ένα νέο σύστημα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, με μια οικονομική διακυβέρνηση. Και έχουν γίνει πολλά και με την ε, οδηγία περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Γι' αυτό και σας ζητώ να με ακούσετε. Όπως ε, ζήτησα και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζήτησα και από τα κράτη-μέλη να δεχτούν κάτι τέτοιο. Δηλαδή να καταβληθεί μία προσπάθεια για συμβιβασμό εμείς. Υποβάλαμε μία πρόταση και αρκούμαστε σε αυτήν. Αλλά κοινότητα σημαίνει συμβιβασμός δεν αναφέρουμε απλώς τις θέσεις μας και μένουμε σε αυτές. Θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό. Γίνεται μια παρέμβαση εκτός μικροφώνου που δεν άκουσαν οι διερμηνείς. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παροτρύνει το Συμβούλιο να κινηθεί. Προβάλαμε ένα πλήρες κείμενο συμβιβασμού και θα συνεχίσουμε να ασκούμε φιλική πίεση προς όλους τους εταίρους για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα έχουμε ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Κάρας, για δύο λεπτά. Κύριε Φαν θα ήθελα να σας πω πως σήμερα δεν κρίνουμε τους τελευταίους μήνες ε, κρίνουμε το αποτέλεσμα της συνεδρίασης του Συμβουλίου. Ε, σε ποια εποχή ζούμε, πού βρισκόμαστε. Εγώ ανέμενα μια αυτοκριτική για τις αδυναμίες μας, μεγαλύτερη ειλικρίνεια για τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία, δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία πήγε ο Σάντης στο Στρασβούργο. εξακολουθούμε να προχωράμε όπως όπως αντί να χτυπάμε στο καρφί. Δεν αναμένω πλέον ηγετικό ρόλο από το Συμβούλιο, αλλά το αναμένω από την Κομισιόν. Αυτό το οποίο αναμένω από το Συμβούλιο είναι να μην καθυστερεί και να μην μπλοκάρει και να στηρίζει την Κομισιόν. Και όταν κάνει ανακοινώσεις να ακολουθούν γρήγορα πράξεις. Επίσης, η νέα αυτή μέθοδος των επιστολών. Δεν μου λέει τίποτα. Λαμβάνουμε γράμματα από τη Μέρκελ και τον Σαρκοζή 24 ώρες πριν τη Σύνοδο. Τώρα λαμβάνουμε επιστολή από τον Μπαρόζο και τον Φαν που απευθύνεται στον εαυτό τους. Επιστολή από τον Ομπάμα, μια επιστολή από τον Καναδά. Θέμε συγκεκριμένα δεδομένα και έργα. Γράψτε λιγότερες επιστολές και αναλάβετε συγκεκριμένες ημερομηνίες για τις πρωτοβουλίες σας. Ευρώπη 2020. Κάντε τη στρατηγική αυτή ένα μέσο και ένα συγκεκριμένο έργο ανάπτυξης και ε, θέσεων εργασίας. Ο, η εισφορά των τραπεζών δεν έχει αποφασιστεί συγκεκριμένα. Ο φόρος των συναλλαγών δεν υπάρχει τίποτα το ευρωπαϊκό. Η εποπτεία των χρηματαγορών μπλοκάρεται στον τριμερή διάλογο. Hedge funds, το ίδιο. CD το ίδιο. Και στη Βασιλεία, και τελειώνω, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή υποστηρίζουν τι πράγμα, μία, έναν ορισμό της οδηγίας ε, κεφαλιακής επάρκειας που δίνει προτερήματα Αμερικάνου Αμερικάνους έναν της Ευρώπης. Η κυρία Μπερές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευτυχώς η στρατηγική 2020 ασχολήθηκε και με την ε, καταπολέμηση της φτώχειας. Φοβούμεθα όμως ότι η στρατηγική δημοσιονομικής ολοκλήρωσης πάει πολύ μακριά και δεν μειώνεται αρκετά η φτώχεια, διότι υποβαθμίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες. Σε σχέση με την οικονομική διακυβέρνηση δεν θα ήθελα να επικρίνω. Θα πρέπει να γίνει μια επικοδομητική συζήτηση και εδώ θα, ήθελα, θα θέλαμε και εμείς να υποβάλουμε ορισμένες προτάσεις. Καταρχήν, ως προς τα μακροοικονομικά ζητήματα υπάρχουν μίζωνες ανισορροπίες και φοβούμεθα το εξής ότι προβάλλουμε το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης σαν να ήταν ύψιστο αγαθό και δεν μιλάμε για τη μέθοδο και τη δυνατότητα μείωσης αυτών των ανισορροπιών που υποβαθμίζουν την Ευρωζώνη και επιτρέπουν στη Citigroup να μην θεωρεί την Ευρωζώνη ως σύνολο. Επίσης, ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι οι κυρώσεις. Δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις μόνο ως προς το έλλειμμα. Θα πρέπει να υπάρχουν και ευφύς κυρώσεις. Εάν ένα κράτος βρίσκεται σε δυσκολίες θα μπορούσαμε να του ζητήσουμε αύξηση των φόρων. Ε, με συγχωρείτε, θα πρέπει να σας διακόψω, λέει ο πρόεδρος. Γκουλάρ, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Ακούσατε το τι είπε ο πρόεδρος της BP που είπε Θέλω τη ζωή μου όπως ήταν πριν. Νομίζω ότι υπάρχουν ε, κυβερνήσεις που εθελοτυφλούν. Δηλαδή θεωρούν ότι δεν υπάρχει κρίση και η ζωή τους κυλάει όπως πριν. Όμως συνέβησαν πολλά. Και έτσι τι κάνουμε. Έχουμε ένα αρχικό σχέδιο Λαροζιέρ το οποίο έχει απαλυνθεί, έχει διαλυθεί και όλοι αντιδρούμε σαν επρόκειτο για μια πολύ μικρή εμβέλεια κρίση. Θα ήθελα όμως ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Το Δεκέμβριο του 2009 το ΕΚΟΦΗΝ μπλόκαρε κάθε δυνατότητα συζήτησης με συναπόφαση. Και Είχαμε πει τότε από την ΕΚΟΝ ότι δεν, θα δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και στις 10 Μαΐου ψηφίστηκε μία εντελώς διαφορετική έκθεση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε επανάληψη ενό τέτοιου σενάριου. Θέλουμε θεσμούς που να λειτουργήσουν από την 1η 2011, αλλά θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που να μην βασίζεται στην καλή θέληση των κρατών και να δίνουν δικαίωμα αρνησικυρίας στα κράτη τα οποία δεν επιθυμούν χρηματοπιστωτική εποπτεία. Δεν μπορούμε δηλαδή να δεχτούμε λύσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Κοζόσνικ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε καλέσει κάποιες φορές τον ε, Επιτρόπο Έχουμε ε, τον κύριο Μόντι και έχει εκπονηθεί και έκθεση Μόντι. Πρέπει όμως οι Ευρωπαίοι να δείξουν τόλμη. Και οι Ευρωπαίοι ηγέτες αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Αυτές οι ελκυστικές ιδέες δηλαδή που διατυπώνονται να τις μετατρέψουν σε έργα, σε πράξεις. Έχουμε ακούσει κάποιες φήμες ότι τόσο και στην Επιτροπή όσο και στο Συμβούλιο υπάρχει η τάση ενός μεγάλου ευρώ και ενός μικρού ευρώ. Είχαμε κάποιες εμπειρίες εμείς με το δυτικό και το ανατολικό Μάρκο, το οποίο υπήρχε κατά το, την περίοδο ψυχρού πολέμου. Και εντάξει, δεν, ήταν και τόσο, δεν είμαι και τόσο αντίθετο. Ο κύριο Πόρτα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν σε σχέση με τον τραπεζικό φόρο και το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θα προτιμούσα λιγότερα λόγια και περισσότερα έργα και δυνατότητες ε, διαπραγμάτευσης, γιατί θα δείτε τι θα γίνει στους G20. Είμαστε σκαπανείς, αλλά σκαπανείς άνευ έργου και άνευ ερίσματος. Πώς μπορείτε να πείτε ότι θέλετε να μειώσετε την φτώχεια στην Ευρώπη και στον κόσμο όταν παντού σε όλους τους εθνικούς προϋπολογισμούς υπάρχουν ε, πολιτικές δραστικής μείωσης των ε, δημοσίων επενδύσεων και των κοινωνικών επενδύσεων. Πώς μπορείτε να υποστηρίζετε την ανάγκη μιας βιώσιμης ανάπτυξης εάν στο μεταξύ όλες οι εθνικές πολιτικές έχουν ένα στόχο αποκλειστικά την μείωση των μισθών και την αύξηση των φόρων, ιδιαίτερα του ΦΠΑ. Γι' αυτό αντιμετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα με το Συμβούλιο. Είναι σαν ένα Βατικανό, όπως έλεγε ο Ζωζέ Σαραμάγκο. Δηλαδή είναι ένα ορθόδοξο Βατικανό, αν μπορούμε να πούμε, που δεν ξεχνά τίποτα αλλά δεν μαθαίνει τίποτα. Έτσι έλεγε ο εθνικός μας συγγραφέας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι όπως είπε ο κύριος Βαν Ρομπόη, μίλησε για προληπτικές κυρώσεις στα δημόσια δημοσιονομικά. Πώς μπορεί να υπάρχουν προληπτικές ε, ε κυρώσεις. Διακόπτει ο πρόεδρος. Πάσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Φανρόμπο, κύριε Μπαρόσο. Στο σημείο 11 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου γίνεται λόγος για την ενίσχυση των προληπτικών μέσων για την επίτευξη των στόχων του Συμφώνου Σταθερότητας. Και μετά από την δημοσίευσή τους ξεκίνησε μία συζήτηση για το τι κάνουν οι διάφορες χώρες και το πώς είναι υποχρεωμένες να επιτύχουν αυτούς τους ε, στόχους και προτάθηκε οι υπουργοί εκείνοι οι οποίοι έχουν οι χώρες εκείνες οι οποίες ε, έχουν ε, τα υψηλότερα ενεργητικά θα βρεθούν να έχουν ένα μειονέκτημα και θα πρέπει να υπάρξει μια κλίδα με βάση την οποία θα λαμβάνονται οι αποφάσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίση, ανοιχτό ζήτημα είναι το πώ θα υπάρξει κάποια αλληλεγγύη στο μηχανισμό σταθερότητα, καθώ ε, φαίνεται πω οι φτωχέ ε, χώρε ε, θα εξακολουθήσουν να χρεώνονται για να διατηρηθεί το επίπεδο των πλουσιότερων χωρών. Δεν είμαι σίγουρο αν αυτό είναι το σωστό. Κύριο Γκρίφιν, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η στρατηγική τη Ένωση για τι Δουλειέ ακούγεται καλή, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Να πάρουμε ένα σοκαριστικό παράδειγμα. Η συμφωνία εμπορίου με την Ινδία η οποία έρχεται θα έχει καταστροφικό αποτέλεσμα στην Ινδική γεωργία και φαρμακοβιομηχανία και δικαίω ανησυχούν οι Ινδοί. Όταν δίνουν τόσα πολλά οι Ινδοί, αναρωτιόμαστε τι κερδίζουν οι μεγάλες Ινδικέ επιχειρήσεις και τι θα κοστίσει στου εργαζόμενους στη Βρετανία και την Ευρώπη. Η απάντηση είναι η μετανάστευση που πλέον δεν θα έχει καθόλου εθνικά όρια και πολυεθνικές επιχειρήσεις θα έχουν αυτόματο δικαίωμα να φέρνουν ε, Ινδού εργάτε, να αντικαταστήσουν π.χ. ειδικευμένου βρετανού εργάτε παραδείγματο χάρη σε χαλιβουργίες και αυτοκινητοβιομηχανίε. Έτσι θα υπονομευθούν οι μισθοί και οι σε εκατοντάδων χιλιάδων Βρετανικών ε, επιχειρήσεων. Πρόκειται για ξεπούλημα στην απληστία των ε, επιχειρήσεων. Γκαρσία Μαρκάγιο. Για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Η χρηματοπιστωτική εποπτεία είναι ε, το μόνο συγκεκριμένο ε, στοιχείο αυτή τη περίεργη ιδέα που ονομάζουμε οικονομική διακυβέρνηση. Και πρέπει να σα πω ότι ουσιαστικά εδώ βρισκόμαστε εν πλήρη συγχύση. Σήμερα το πρωί μα είπε ο πρόεδρο ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία, μα είπε ότι πρέπει να ε, κινηθούμε. αλλά αυτό ουσιαστικά είναι σαν ε, να κάνουμε οικονομίες στην αλήθεια. Ούτε ε, μπορούμε να κινηθούμε, αν, ε, όχι προς την κατέστη που θα σας πω εγώ, ούτε και το άλλο που μας είπε ισχύει. Η συμφωνία που μας αναφέρει το Συμβούλιο είναι μια συμφωνία των ελαχίστων, που θέλει κάποιες αρχές που θα έχουν ως μόνο καθήκον να προτείνουν κάποια τεχνικά πρότυπα εναρμόνισης ε, για ομοιόμορφη ερμηνεία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Δεν χρειάζεται τίποτε να κάνουμε με το 290 άρθρο, το έχει πει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το οποίο λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το εξή. Πρώτον, ότι οι πανευρωπαϊκές τράπεζες πρέπει να εποπτεύονται από μία ευρωπαϊκή αμυγός αρχή, η οποία θα υπόκειται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και κάποιε τράπεζε, οι οποίε όταν χρεοκοπούν μπορούν να μα παρασύρουν όλου, θα πρέπει να είναι υπό εποπτεία και επιτήρηση. Όταν μια από αυτέ τι τράπεζε μπαίνει σε δυσκολίε, η τραπεζική αρχή να έχει μια εργαλειοθήκη για να μην υπάρξει μετάδοση αυτού του προβλήματο, ε, για να γίνει η σωστή εκαθάριση και να μην ε, ε, πληγούν οι φορολογούμενοι. Και Επίσης να υπάρχουν δύο ταμεία τα οποία χρηματοδοτούνται από τον ίδιο κλάδο με βάση και την αρχή ορυπαίνων πληρώνει ώστε όταν κάποιος ε, κάνει κάποιες υπερβολές όπως χαριτολογώντας έχουν πει κάποιοι να μην πληρώνουν οι υπόλοιποι φορολογούμενοι. Πριν αρχίσει η Ισπανική Προεδρία σας δω... Δυστυχώς έχετε υπερβεί το χρόνο σας. Ο Μάικλ Κάσμαν, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπαρόζο, κύριε Φωνορόμ έχω 90 δευτερόλεπτα, δεν είναι και πολύς χρόνο, αλλά θα ήθελα να σκεφτείτε εσεί και το Κοινοβούλιο το εξή για την ε, μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση των στόχων της χιλιετίας λέει ο εισηγητής ότι τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν ότι σε 90 δευτερόλεπτα μέχρι να κάτσω κάτω δηλαδή 45 ε, άτομα θα έχουν ε, πεθάνει κάθε, δηλαδή ένας κάθε δύο δευτερόλεπτα στον αναπτυσσόμενο κόσμο θα έχουν πεθάνει από επιπλοκές στη γέννα από διάφορες μεταδόμενες νόσους από το AIDS, από την υπατήτηδα από την φυματίωση, από την ελονοσία κάθε ε, δευτερόλεπτο, δύο δευτερόλεπτα μάλλον, ένα θάνατο. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να εκπληρωθούν οι δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει για του ε, αναπτυξιακού στόχου τη χιλιετία σε επίπεδο G20, αλλά και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Και εμεί, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε αυτά τα ζωτική σημασία σχέδια στι αναπτυσσόμενε χώρε. Μου μένουν 20 δευτερόλεπτα και θα σας ε, παρακαλέσω να δείξετε υπομονή. Ε, να μην μιλήσουμε κανείς, να μην μιλήσει κανείς αυτά τα λίγα, λεπτά που, τα λίγα δευτερόλεπτα που μου απομένουν, αλλά να σκεφτούμε λίγο αυτούς τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους αυτά τα 90 δευτερόλεπτα. Thank you, ε, Ευχαριστώ η κυρία Μπόουλς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Φαν Ρομπο, χαίρομαι που σας βλέπω εδώ πέρα και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών θα ήθελα να σας βλέπω περισσότερο στην Επιτροπή ως επικεφαλής της Task Force γιατί όταν ε, έχετε ιδέε οποιαδήποτε πολυμερή εποπτεία θα έρχεται σε εμά υπό την απόφαση και όσο δεν μα ενημερώνετε τόσο περισσότερο χρόνο θα χρειαστούμε να κατανοήσουμε τι αποφάσει και έχουμε και εμεί κάποιε ιδέε. Για να έρθω τώρα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, βλέπω πώς ζητούν γρήγορη δράση στο πακέτο επαπτείας, στο ΕΕΦΜ και στα παράγωγα. Δεν ε, δε τονίζεται εδώ πέρα η τρίτη οδηγία κεφαλιακών ε, απαιτήσεων. Κάτι το οποίο βεβαίως έγινε υπό την πίεση των τραπεζών ήδη πριν από την ε, τράπεζα και έτσι γίνεται ελκυστική αυτή η κερδοσκοπική δραστηριότητα η οποία ξεκίνησε την κρίση. Η αυτή, η τρίτη οδηγία, αυτομάτως θα περιόριζε το τραπεζικό καζίνο χωρίς να χρειάζεται να πειράξουμε τις τράπεζες. Γιατί λοιπόν δεν είναι το πρώτο κομμάτι της εφαρμογής. Τέλος, ε, υποστηρίζω το να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα του τεστ κοπόσεων των τραπεζών. Έχουμε αργήσει τουλάχιστον κατά ένα χρόνο και ίσω θα είχαμε λιγότερα προβλήματα με το δημόσιο χρέο αν είχε γίνει νωρίτερο. Πρέπει να γίνουν, εν περιπτώσει, τώρα και να καλύπτουν όλε τι ανησυχίε των τραπεζών. Αλλιώ θα γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Ευχαριστώ η κυρία Νίκη Τζαβέλα για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, είναι τιμή μας και χαρά μας να σας βλέπουμε, γιατί τους άλλους δύο ε, Προέδρους τους βλέπουμε και στο Στρασβούργο και θα ήθελα να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι η νυφάλια προσέγγισή σας στα θέματα αυτή την περίοδο ήταν πολύτιμη. Κύριε Πρόεδρε, στο τελευταίο Συμβούλιο η Γερμανία δέχτηκε ότι η ένωση χρειάζεται κάποιας μορφής οικονομική διακυβέρνηση. αρνήθηκε όμως να αποδεχθεί την εύλογη εισήγηση της γαλλίας ότι η διακυβέρνηση αυτή πρέπει να ασκείται στο επίπεδο των 16 της ευρωζώνης τουλάχιστον για την αρχή. έτσι οδηγούμαστε στη διαμόρφωση οικονομικής διακυβέρνησης των 27 και σας ερωτώ τι είδους κοινή οικονομική πολιτική μπορεί να ασκήσουν 27 χώρες με 18 διαφορετικά νομίσματα, διαφορετική φορολογία, διαφορετικό ύψος ε, επιτοκίων δανεισμού κλπ. Φοβάμαι μήπως οδεύουμε πάλι στην προβληματική δομή της ε, Ευρωζώνης. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Ερενχάουζερ για ένα λεπτό. Σύντομα, λίγα λόγια για την Ευρώπη 2020. Θεωρώ πως μπορούμε να μιλάμε για πρόοδο όταν ο στόχος είναι η περισσότερη ανάπτυξη και η φορεία, αλλά βεβαίως δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα. Το βασικό ζήτημα είναι πως θα φύγουμε από αυτή τη μανία για ανάπτυξη, πώς θα εμποδιστούν αυτές οι κρίσεις στο μέλλον. Και αν θέσουμε αυτό το ερώτημα, δεν μπορούμε παρά να οδηγηθούμε σε θεμελιώδη μεταρρύθμιση του χρήματο ψηφιακού ε, συστήματος. Μήπως θα έπρεπε να ξαναέρθει στα χέρια του κράτους η δημιουργία του χρήματος πράγματα όμως και ερωτήματα τα οποία ε, απαιτούν μια ισχυρή και ανεξάρτητη πολιτική. Ευχαριστώ. Χίπνερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι οι φορολογικές και χρηματοοικονομικές μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μια πολιτική ανάπτυξης. Γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω για την ε, πολιτική συνοχής μέσα στα πλαίσια του Μηχανισμού Ευρώπη 2020. Στα συμπεράσματα το Συμβούλιο μας μίλησε για μια πολιτική συνοχής που να εντάσσεται στην Ευρώπη 2020 ήταν και το μόνο θετικό μήνυμα από τη στρατηγική της Λισαβόνας μετά από την ανακοίνωση του Μαρτίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό διότι τίθενται δεσμευτικοί στόχοι για μεταφορά πόρων προς ε, ένα κράτος μέλος ή περιφέρεια ή πόλη έτσι ώστε οι περιφέρειες να μετατρέψουν τους κοινούς στόχους σε μία δική τους πραγματικότητα. Επίσης να επιτύχουμε απτούς στόχους και υπάρχει και ένας αποδοτικός ε, μηχανισμός κυρώσεων. Για την οικονομική διακυβέρνηση υποστηρίζω το ότι θα πρέπει να κινηθούμε πέρα από την φορολογική εποπτεία και να καταπολεμήσουμε τις αδυναμίες και τις ανισορροπίες. Και θα πρέπει να πούμε σήμερα με δυνατή φωνή γιατί δεν ε, λειτουργήσε η φορολογική εποπτεία και γιατί δεν απέδωσε το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Ίσως στα πλαίσια της φορολογικής πειθαρχίας να φτάσουμε μια καλύτερη ε, διαχείριση αλλά όχι μια πραγματική οικονομική διακυβέρνηση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χαράγουι Ατόντο, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε, κύριε Βαν και Μπαρόσο. Σημερίζομαι μέσα στο το εξής. Στην συνάντηση την Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε σημαντικές αποφάσεις που ήταν αδιανόητες τέσσερις μήνες πριν και θα πρέπει να είμαστε θαραλέοι και να το παραδεχτούμε. Νομίζω ότι ότι οι κρίσεις οδηγούν την Ευρώπη προς τα εμπρός. Αυτό κατέδειξε και η ιστορία. Και έτσι έχουμε μία σειρά αποφάσεων, βήματα δηλαδή που είναι πολύ σημαντικά για την οικονομική οικοδόμηση. Βεβαίως μία από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όχι ίσονος ήταν η μεταρρύθμιση της ε, συνθήκης και να συγκληθεί μια διακυβερνητική για να ανανεωθεί το πρωτόκολλο 36 της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό σημαίνει ότι θα ενσωματωθούν ε, άλλοι 18 βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι θα υπάρχει καλύτερη εκπροσώπηση σε σχέση με αυτή που είχαμε μέχρι τώρα. Σε αυτά τα πλαίσια θα ήθελα να τονίσω την σημασία του γεγονότος ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δέχτηκε να διευρύνει την εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σήμερα η διακυβερνητική ήδη έλαβε αυτή την απόφαση σε επίπεδο 27 και σας συγχαίρω κύριε Βαν Ρομπόη για αυτή την απόφαση γιατί θα πρέπει να επιταχυνθεί η κύρωση από τα 27 κοινοβούλια έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει σωστότερη εκπροσώπηση με 18 επιπλέον βουλευτές που θα μπορέσουν να εκπροσωπήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Πρέντα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φαν και κύριε Μπαρόζο. Πρώτα απ' όλα Καλωσορίζω την απόφαση τη προηγούμενη εβδομάδα ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ξεκινήσει διαπραγματεύσει με την Ισλανδία. Σήμερα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου η έκθεσή μου για την προσχώρηση της Ισλανδίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε δεκτή με μεγάλη πλειοψηφία. Οι συνάδελφοί μου είπαν ότι συμφωνούν να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα αυτή. Θα πρέπει ωστόσο να εξευρεθεί μια κοινή λύση σε τομείς όπως είναι η αλληλεία ή η γεωργία. Πιστεύουμε ότι η Ισλανδία μπορεί να πετύχει τους στόχους της, έχει ήδη άλλωστε πετύχει ορισμένους εκφτών και μπορεί να σε το κοινοτικό κεκτημένο και να γίνει ένα νέο μέλος ε, της ευρωπαϊκής οικογένειας. Μπορεί πιστεύω να συμβάλλει διότι έχει δημοκρατική παράδοση, έχει εμπειρία στην ε, προστασία του περιβάλλοντος και μπορεί να εφαρμόσει τις ευρωπαϊκές πολιτικές στην περιοχή της Αρκτικής. Φυσικά και η Ισλανδία θα κερδίσει πράγματα και δεν μιλάμε μόνο για την οικονομική σταθερότητα αλλά και για την μεγαλύτερη επιρροή σε Διεθνέ επίπεδο σε ό,τι αφορά αποφάσει που αφορούν την εσωτερική αγορά. Γνωρίζουμε από την άλλη πλευρά ότι σε ό,τι αφορά την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων ε, στην Ισλανδία. Η κυβέρνηση ξεκίνησε διάλογο. Ε, υποστηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο διάλογος αυτός και ίσως ε, γίνει μια χρήσιμη συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να επιλέξουν με τα λόγου γνώσεως οι Ισλανδοί το αν θέλουν ή όχι η χώρα τους να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο τέλος της διαδικασίας ε, αυτής θα γίνει και δημοψήφισμα στην Ισλανδία για να ε, φανεί τι επιθυμεί ο πληθυσμός της χώρας. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Λαμπρινίδης για 1,5 λεπτό. Τα χρόνια του ευρώ του Νότου και του Βορρά ε, απέκλειναν μεταξύ του αντί για να συγκλίνουν. Ο κύριο λόγο είναι ότι ήταν πολύ διαφορετικά δομημένε. Ο Νότο, υπηρεσίε, αγροτικά, ο τουρισμό, ο Βορρά, βαριά βιομηχανία, εξαγωγέ. Ο Νότο επομένω έπρεπε να αλλάξει διδικά τι δομέ οικονομία του μέσα πολύ λίγα χρόνια. Ανταυτού αναπτύχθηκε μέσω κατανάλωση, μέσω φτηνών δανείων που επέτρεπε το ευρώ, μέσω υπεχρέωση. Ενώ οι βιομηχανικέ χώρε αναπτύχθηκαν επειδή μπορούσαν πλέον να εξάγουν φτηνότερα και ευκολότερα να λοιπόν γιατί και πού απαιτεί το οικονομική διακυβέρνηση. η έλλειψή της επέτεινε τόσο τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα κάποιων κρατών μελών όσο και τα αναπτυξιακά μειονεκτήματα άλλων. για να βγει σήμερα ο νότος αλλά και άλλοι από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης πρέπει να μπορούν εκτός από δημοσιονομικές προσαρμογές να δανείζονται φτηνότερα για να επενδύουν στην ανάπτυξη και να εξάγουν συμπεριλαμβανομένων μέσω ομολόγων ευρωομολόγων. κι όμως ακριβώς τώρα η συγκριτικά πλούσια γερμανία επιδίδεται σε ένα πρόγραμμα των περικοπών τόσο περιορίζοντα την εσωτερική τη κατανάλωση όσο και καθιστώντα τον εαυτό τη πρωτίστω πιο ελκυστικό στι χρηματοπιστωτικέ αγορέ απέναντι στου εταίρου τη. τέτοια μέτρα δεν συνιστούν κοινή ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική. μετατρέπουν δυνητικά τα κράτη μέλη σε στιγνού ανταγωνιστέ για περιορισμένα κονδύλια αντί για σε αλληλέγγυου εταίρου και βάζουν στην ίδια προκρούστια κλίνη των περικοπών επιτείνοντας έτσι πλεονεκτήματα κάποιων και μειονεκτήματα άλλων και βάζοντας κάποια κράτη μέλη σε μια πολύ αρνητική αφετηρία για την επίτευξη των κοινών υποτίθεται στόχων του. 2020. Ευχαριστώ. για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έναντι της ΟΚΕ χρησιμοποίησατε μία εικόνα ε, λέγοντας ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να περισσώσουμε την κατάσταση, ε, κολυμπώντας την απέναντι αχθή. Ακτή, με συγχωρείτε. Αυτό ήταν αδιανόητο για μερικές χώρες και αυτό το γνωρίζω πολύ καλά. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε τις οσίβιες λέμβους νωρίτερα. Θα έπρεπε να τις ε, είχαμε ήδη δημιουργήσει. Και χρειάζεται αυστηρή εποπτεία των εθνικών προϋπολογισμών. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνει. Θα εποπτεύσει τους εθνικούς ε, προϋπολογισμούς πριν εγκριθούν από το κράτος, από τα κράτη. Ο κύριος Όλι Ρεν μίλησε για ε, θάρρος, για θαρετή προσέγγιση, η οποία θα πρέπει όλο ένα και να επιτείνεται. Αλλά εάν μιλάμε για προτεκτοράκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτιμώ αυτό το προτεκτοράτο παρά το προτεκτοράτο τεχνοκρατών. Γιατί πολλοί είπαν ότι δεν ε, τους ενδιαφέρει το ευρώ εφόσον δεν βρίσκονται στην Ευρωζώνη. Εμένα όμως με ενδιαφέρουν τα εθνικά νομίσματα και ας ανήκω στην Ευρωζώνη γιατί αυτό σημαίνει να είμαστε Ευρωπαίοι. Και τέλος, γνωρίζω ότι σε κρίσεις είναι δύσκολο μιλάμε για την καταπολέμηση της φτώχειας αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ε, καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια. Και το έτος 2010 που είναι έτος κατά της φτώχειας να μην αποτελεί μία απλή δήλωση, αλλά να προβάλλουμε έμπρακτα πολιτικές. Ευχαριστούμε. Η κυρία Τράουτμαν, για ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, μας είπατε πριν ότι η θέση των Ευρωπαίων πρέπει να είναι αποφασιστική και ενιαία για να φτάσουμε στην G20 γιατί τίθεται θέμα αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο διεθνές προσκήνιο. Πάνω απ' όλα όμως ε, πρόκειται για την αξιοπιστία της απέναντι στον πολίτη που περιμένει η Ένωση να μπορεί να έχει ένα μέσο, ένα εργαλείο που θα την βγάλει από την κρίση. Πρώτον, περίμενα ε, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου να ε, εξισώνουν τη μακροοικονομική εποπτεία, την ρύθμιση των αγορών με όλα τα άλλα θέματα. Αυτό δεν έγινε. Δεύτερον, αλληλεγγύη. Θα πρέπει και πρέπει να είμαστε ηγέτες, αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα κατασκευαστικό ελάττωμα στην ΟΚΕ. Το ευρώ σήμερα είναι το 25% των παγκόσμιων αποθεματικών ε, της τράπεζας, των κεντρικών τραπεζών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει συντονισμό των οικονομικών ε, πολιτικών σε εθνικό επίπεδο. Το ευρώ δεν θα πρέπει να είναι το σύμβολο ε, μιας ε, δαπανηρής ζωής. Και δεν πρέπει μόνο να καθησυχάσουμε τις αγορές αλλά και τους πολίτες για το ότι είμαστε ικανοί να εξέλθουμε μαζί από την κρίση. Επίσης, ό,τι αφορά τη μεγαλύτερη λιτότητα, ε, αυτό δεν θα πρέπει να οδηγεί σε μεγαλύτερη ύφεση. Χρειαζόμαστε αποδείξεις για το ότι η στρατηγική 2020 θα συνοδεύεται πράγματι από, απαραίτη, από τους επαρκείς πόρους που θα προσανατολίσουν την οικονομία προς τη μελλοντική απασχόληση, μελλοντικές δαπάνες, προς τις ε, ε, την αλληλέγγυα ανάπτυξη. Υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις, ε, μετά μπορεί να υπάρξει οργή, μετά μπορεί να υπάρξει φόβος. Ε, δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει το σύμβολο μιας βίαιης λιτότητας. Ευχαριστώ. Ντελβό για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, συχνά λέμε ότι ανάγκα θεοί και θεοί πείθονται. Πρέπει τώρα να είμαστε όμως και καινοτόμοι και δημιουργικοί. Εξού λοιπόν και χαίρομαι ε, για αυτό το βήμα που ελπίζω να είναι ένα γιγάντιο βήμα προς μια πραγματική οικονομική διακυβέρνηση. Αν και βέβαια ο πραγματικός συντονισμός των οικονομικών πολιτικών μάλλον θα παραμείνει ανεπαρκής. Ε, ε, για να φτάσουμε σε δημοσιονομική ομοσπονδοποίηση δεν θα πρέπει να μας πιέζουν οι συνθήκες αλλά θα πρέπει να το έχουμε αποφασίσει εμείς οι ίδιοι. Χαίρομαι πάντως με την απόφαση του Συμβουλίου για την ενίσχυση της προληπτικής διάστασης ε, του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας. Βέβαια, πραγματική δημοσιονομική πειθαρχία χωρίς κυρώσεις για τους παραβαίνοντες δεν υπάρχει. Αυτά τα ενισχύσατε αλλά δεν τα διευκρινίσατε και λυπάμαι γι' αυτό. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ικανοποίηση μεταξύ άλλων για τις διάφορες κατευθύνσεις όπως αυτό το πίνακα που είπατε αποτελεσμάτων και βαθμολογίας, ε, για τον οδικό χάρτη, για την ανάπτυξη, τη βιώσιμη, για την ανταγωνιστικότητα για το τραπεζικό τώρα φόρο, για το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, για την επιτάχυνση ε, των διαφόρων μεταρρυθμίσεων. Όλες αυτές οι αποφάσεις ε, και προσανατολισμοί, κύριε Πρόεδρε, πριν από κάποιους μήνες, ίσως και κάποιες εβδομάδες, φαίνονταν ανεδαφικές, μη ρεαλιστικές και καθαρά ε, στη σφαίρα της, του υποθετικού. Και έχετε δίκιο ότι πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή κουλτούρας που έχει γίνει τελικά μετά από μικρά μεταλλά. Τώρα υποχρεωτικά πια τον Οκτώβριο τα κράτη θα πρέπει πολύ συγκεκριμένα να κάνουν πράξη αυτές τις ε, κατευθύνσεις. Και εκεί θα δούμε αν πρόκειται για ένα γιγαντιαίο ιστορικό άλμα από πλευρά Συμβουλίου ή για ευσεβεί πόθους. Κάτι το οποίο θα ε, μα ε, λυπήσει όλου και δει ε, του πολίτε που θα υπομείνουν τη συνέπεια ε, της αποτυχίας στην καθημερινή του Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τζιάν Λούκα Σούστα, για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, επειδή είμαι μεταξύ των τελευταίων που θα λάβουν το λόγο, θα ήθελα να σας ενθαρρύνω. Υπενθυμίσατε ότι δεν εκφράζετε τις κυβερνήσεις αλλά την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο είναι αυταπόδεικτο αλλά φαίνεται ότι δεν είναι για πολλούς. Θα θέλαμε λοιπόν να επιμείνετε στο ρόλο σας έτσι ώστε η σταθερή προεδρία να επιβάλλει στις κυβερνήσεις να περάσουν από τα λόγια στις πράξεις. Εκτιμούμε το έργο σας τους τελευταίους μήνες στη δημιουργία της Task Force και το γεγονός ότι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων υπέγραψαν ένα συγκεκριμένο έγγραφο, διότι αν όλα αυτά μεταφραστούν σε πραγματικότητα θα είναι κάτι το εκπληκτικό. Βεβαίως δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα υπάρξει πραγματικά φόρος τραπεζικών συναλλαγών. Κατά πόσο δηλαδή θα υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Ας δούμε τα συμπεράσματα της Task Force για να δούμε κατά πόσο η οικονομική διακυβέρνηση θα αποτελέσει πραγματικότητα. Φτάσαμε στη συνθήκη της ε, Λισαβόνας και φτάσαμε σε μια μεγάλη καινοτομία. Ας ελπίσουμε ότι η σταθερή Προεδρία θα οδηγήσει στην υλοποίηση αυτών των στόχων. Ευχαριστώ, Χεκμαρκ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτά που μας είπατε σήμερα. Νομίζω πως όλοι καθα... καλωσορίζουμε τα συμπεράσματα και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τρία πράγματα θα ήθελα να σχολιάσω. Πρώτα απ' όλα για το ευρώ. Νομίζω πως αν επιτυχάνουμε αυτά τα πράγματα που έχουμε με αυτόματες κυρώσεις και προβλέψιμες για όσους δεν ακολουθούν τους κανόνες θα έχουμε ένα πιο ισχυρό πλαίσιο και ίσως να δούμε την αναγέννηση του ευρώ σε πολύ ισχυρότερο πλαίσιο από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Αυτή θα είναι η συνεισφορά στο μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτό όμως σημαίνει πως πρέπει να κάνουμε και πολλά πράγματα για την ανάπτυξη. Καλώς ορίζω τους σαφείς στόχους που έχουν τεθεί, αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους πως ε, σκληρή δουλειά και οι δύσκολες επιλογές πρέπει να γίνουν. Δεν γίνονται με το να θέτουμε απλώς στόχους, το μάθαμε αυτό από τη Λισαβόνα πρέπει να μπορούμε να λαμβάνουμε τις δύσκολες αποφάσεις να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για περισσότερο εμπόριο, επενδύσεις και καινοτομία. Αυτά πρέπει να γίνουν, αλλιώς μόνο λίγο χρόνο κερδίσαμε και θα επανέλθουν τα ίδια προβλήματα. Τέλος, περνάμε τώρα σε μια φάση παγκόσμιας οικονομίας που θα χαρακτηριστεί από τη μείωση ελλημάτων και στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη και όλοι ξέρουμε τους κινδύνους με την συστολή αυτή της οικονομίας. Πρέπει ταυτόχρονα να κινητοποιηθεί η οικονομία και υπ' αυτή την έννοια αυτά τα οποία έχουν αναφερθεί για το γύρο του Ντόχας πρέπει να ενισχυθούν κατά τρόπον ώστε να είναι συνεκτικά. Δεν αντιλαμβάνομαι τον φόρο στις συναλλαγές που θα εμποδίσει το εμπόριο και τη ρευστότητα και θα βλάψει τις φτωχές χώρες με λύματα. Έτσι, κύριε Πρόεδρε, θα κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, κύριο Ζαλεύσκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν και του Συμβουλίου, η κρίση μας έδειξε πως ε, δεν είμαστε ακόμα αρκετά ενωμένοι παρά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν έχουμε ακόμα πραγματική οικονομική διακυβέρνηση. Θα πρέπει λοιπόν να υψώσουμε τα ανάστημά μας. Είχαμε αυτό το φαινόμενο ντόμινο, είχαμε κρίση σε μια χώρα που επεκτάθηκε. Καλώς ορίζω τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Νομίζω πως υπάρχει ανάγκη οικονομικού συντονισμού πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις για τις χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες και χαίρομαι επίσης για το ότι δεν δημιουργήσαμε ένα αποκλειστικό κλαμπ για τα μέλη Ευρώ-ΣΥΝ. Το ευρώ είναι ένα νόμισμα για αυτούς που είναι ήδη μέσα αλλά και για όσους θέλουν να μπουν. Και νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να αφήσουμε την πόρτα ανοιχτή για τις χώρες εκείνες που θα μπουν στο μέλλον και θα πρέπει να λάβουμε μέρο και στην διαδικασία λήψη αποφάσεων. Γιούτα Στάνικο. Κύριοι Πρόεδροι, είναι καλό να προσπαθήσουμε όλοι να παραμερίσουμε τις αιτίες κρίσεις και να στοχεύσουμε σε ανάπτυξη και δουλειές, αλλά να μάθουμε και από τα λάθη του παρελθόντος και δεν πρέπει να χάσουμε το στόχο από τα μάτια μας στην καταπολέμηση της φτώχειας και είναι κρίμα το ότι οι αρχηγοί των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων δεν ήταν διατεθειμένοι να ευθύσουν τις προτάσεις της Κομισιόν για την καταπολέμηση της φτώχειας. Τέλος, το μήνυμα του Συμβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα είναι πως δεν ασχολείται με τους στοχούς η Ευρώπη. Βελτιώθηκαν οι αρχικοί στόχοι και έμειναν τρία νούμερα και η μείωση των φτωχών κατά 20 εκατομμύρια. Αυτό είναι πάρα πολύ λίγο. Και θα επιθυμούσαμε να μειωθεί η φτώχεια κατά 25%. Γιατί τελικά η φτώχεια είναι κίνδυνος για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Η κυρία Ιζαμπέλ τώρα. Καταρχήν θα ήθελα να αποτανθώ στον κύριο Πανρομπόη, ο οποίος μόλις αποχώρησε. Θα ήθελα όμως να πω προς εκείνον και προς όλους ότι ε, δεν πρόκειται για διακομόδηση διότι ε, πολλοί από μας είμαστε οι καλύτεροι σύμμαχοί του σε θέματα ελέγχου του προϋπολογισμού και αποτείνομαι σε εσά κύριε Μπαρόζο έγινε λόγο στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για μια νέα ε, διακυβερνητική συνέλευση έτσι ώστε όλοι να υπόκεινται στους ίδιους ε, δημοσιονομικούς κανόνες ελέγχου κυρίως έτσι ώστε να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ ευρωπαϊκών δαπανών και εθνικών δαπανών έτσι ώστε να υπάρχει ένας σωστός μηχανισμός εποπτείας και κυρώσεων. Ρώση. Άκουσα με ενδιαφέρον τα σχόλια της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Μίλησαν για στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Οικονομική Διακυβέρνηση για την Ευρώπη 2020. Η Task Force το Σεπτέμβριο θα τελειώσει με τις εργασίες της και θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις. Θα υπάρξουν προτάσεις και στον τομέα του περιβάλλοντος. Ζούμε σε μια Ευρώπη η οποία διανύει μια πολύ μεγάλη περίοδο κρίσης θεωρούμε ότι μέχρι το 2020 θα πρέπει να δημιουργηθούν 8 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας που θα αφορά μία ε, διαδικασία εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θέλουμε να προετοιμάσουμε τις νέες γενναίες για μία νέα Ευρώπη. Ο κύριος Μάριο Μάουρο. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, ο κύριος Βανορομπόη, μίλησε για, χρησιμοποίησε μία λέξη, βαθμιαία. Βαθμιαία σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε και το βαθμό ή διαβάθμιση θέλησης των κρατών μελών και άρα τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να συμπληρωθούν. Πώς μπορούμε να περάσουμε από το βαθμιαίο στο ταχαίος, πώς μπορούμε να περάσουμε στο καλύτερο και τάχιστα, διότι η πολιτική ηγεσία αυτή τη στιγμή είναι ελληματική. Προσπαθούμε να υλοποιήσουμε πρωτοβουλίες, αλλά θα πρέπει να είναι μία ηγεσία που να προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία να μπορέσει πραγματικά με προτάσεις πρωτοβουλίας να καινοτομήσει. Κύριε Παρόζο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, κάποιοι που έθεσαν ερωτήσεις έφυγαν. Εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να απαντήσω. Πρώτα απ' όλα για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Στρατηγική 2020 που ενισχύει πολλά την κυρία Κορίν Βόρτμαν ε, Κόλ η οποία έχει αγωνιστεί για τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στρατηγική αυτή. Νομίζω πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να παίξει ένα ρόλο κλειδί. Είναι η κοινή μας ευθύνη για να οδηγηθούμε ξανά σε ανάπτυξη και θέσεις εργασία ε, για να μην επαναλάβουμε τα όσα έγιναν την τελευταία δεκαετία. Επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το ρόλο του συνομοθέτη για την νομοθεσία αυτή για τις πέντε κύριες πρωτοβουλίες. Ξεκινήσαμε με την ψηφιακή ατζέντα και θα ακολουθήσουν έξι ακόμα πριν το τέλος του 2010. Μιλάμε για ένα εντατικό πρόγραμμα θα έχουμε και μια σειρά νομοθετικών προτάσεων και βασιζόμαστε στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να περάσει την νομοθεσία γρήγορα. Αναμένω δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να, κινη... για να εγκριθούν γρήγορα αυτές οι πρωτοβουλίες. Δεύτερον, θεωρώ πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει ένα πολύ πιο ενεργό ρόλο υπό τη στρατηγική της Λισαβόνας για να ορίσει τη στρατηγική 2020 ε, λαμβάνοντας θέσεις έγκαιρα και προληπτικά. Επίσης θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο στην κινητοποίηση των εθνικών κοινοβουλίων, αλλά νομίζω πως τώρα υπάρχει περιθώριο για να φύγει αυτός ο διάλογος από τη γενική συζήτηση, τη γενική συζήτηση που, στην οποία καμιά φορά και εγώ συμμετείχα στην πρώτη φάση, και να πάμε προς πολύ πιο συγκεκριμένα ζητήματα όπως οι πέντε βασικοί στόχοι της στρατηγικής απασχόληση, έρευνα και ανάπτυξη, ενέργεια, εκπαίδευση και καταπολέμηση της φτώχειας. Τα εθνικά κοινοβούλια θα παρακολουθούν το πώς οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν σωστά τους εθνικούς στόχους για την Ευρώπη 2020 και τις συστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρω πως κάποιοι δεν είστε ικανοποιημένοι, θα προτιμούσατε πιο φιλόδοξους στόχους όσον αφορά την παρακολούθηση της στρατηγικής, αλλά υπάρχουν βελτιώσεις εδώ πέρα και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην υποτιμάτε ε, το δυναμικό του. στόχου. θα υπάρχουν τώρα εθνικά προγράμματα και συγκεκριμένοι εθνικοί στόχοι καθιστά δυνατόν να επιτηρούμε με συγκεκριμένο τρόπο όχι μόνο το τι γίνεται αλλά ποια χώρα κάνει τι σε όλους αυτούς τους στόχους. Και αυτό πρέπει να γίνει από το Κοινοβούλιο με τα άλλα όργανα. Πρώτη προτεραιότητα είναι η φτώχεια και πρέπει να εκμεταλλευτούμε το ευρωπαϊκό του καταπολέμηση τη ε, φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού για να ξεκινήσουμε αυτέ τι πολιτικέ. Δεν ήταν εύκολο να συμφωνήσουμε σε στόχο. Κάποιοι είχαν αμφιβολίε όσον αφορά την επικουρικότητα και όμως καταφέραμε να ε, αποσπάσουμε κάποια δέσμευση και πρέπει αυτό να το κάνουμε ήδη ορατό από φέτος γιατί είναι ε, έκτακτη η κατάσταση και στο κοινωνικό μέτωπο. Τέλος, για να επανέλθω στο στόχο της Ευρώπης 2020, ως αρχή του προπολογισμού πρέπει να παίξει και ένα ρόλο για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρέπει να οριστούν λοιπόν οι στρατηγικές αυτές. Θα έρθουμε με την αναθεώρηση του προπολογισμού τον Σεπτέμβριο και τότε θα είναι η στιγμή να ξεκινήσει μια ευρεία συζήτηση για το τι θα γίνει με τις δημοσιονομικές πρακτικές και κάποιες ιδέες που προτάθηκαν στην ε, προκατακτική συζήτηση με το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω το έγγραφο Λάμασουρ που παρουσιάστηκε στην εβδομάδα, πρέπει αυτή την εβδομάδα, για το πώς θα χρηματοδοτηθεί ε, σε καιρό κρίσης η Ευρώπη 2020 και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε τι θα ξοδευτεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο είναι κάτι που θα το αποφασίσει το Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα. Να σα πω εκ μέρου τη Κομισιόν πω εμεί οπωσδήποτε θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σα. Κάτι άλλο που ακούστηκε από τον κύριο Κάσμαν αφορούσε του στόχου τη χιλιετία. Συμφωνώ πλήρω με όλα όσα είπε και με την ανάγκη να παραμείνει μια ορμή σε αυτό το ζήτημα, ειδικά τώρα που πιέζονται οι προπολογισμοί των κρατών μελών. Θα είναι δύσκολο οπωσδήποτε και μάλιστα ε, ως προς αυτό είναι καλά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και στην επιστολή μαζί με τον πρόεδρο Φαν Ρόμποϊ που απίθυνα στους αδέλφους των G20 το αναφέρουμε. Επαναβεβαιώνουμε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις δεσμεύσεις των κρατών μελών και λέμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους στόχους αυτούς μέχρι το 2015. Καλό θα ήταν να κάνουν και όλοι Αυτά θα πούμε στους G20 και στους G8 ε, το Σαββατοκύριακο αυτό στον Καναδά. Κάποιοι ρωτήσετε και για τα τεστ αυτά κοπόσεως των τραπεζών. Ήταν μια θετική ανακοίνωση πριν από την σύνοδο του Τορόντο, τον G20, για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στις ευρωπαϊκές τράπεζες και τις πρόπτικες. Το πώς ακριβώς βεβαίως θα γίνει το συζητάμε τώρα με όλους τους ενδιαφερομένους και συγκεκριμένα με την Επιτροπή ε, Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Τραπεζικών Αρχών με τους ε, αντίστοιχους ε, χρηματοπιστωτικούς επόπτες και νομίζω ότι όπως γνωρίζετε η απόφαση θα ληφθεί τις επόμενες ημέρες. Θα πρέπει να υπερασπιστούμε αυτή την προσέγγιση έτσι ώστε να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό δείγμα λαμβάνοντας υπόψη την χρονική πλαισίωση ε, δημοσίευση των αποτελεσμάτων, δηλαδή τον Ιούλιο. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, πιο πρόσφατες αλλαγές σε σχέση με το δημόσιο χρέος. Θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τις ε, πρόσφατες πιέσεις που δέχτηκαν τα δημόσια, δημοσιονομικά και οι εθνικοί προϋπολογισμοί και νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει και το δημόσιο χρέος γενικότερα και πιστεύω ότι θα ληφθούν αποφάσεις τις επόμενες ημέρες. Μερικοί αναφέρθηκαν και στο θέμα της ε, διαρροής στον κόλπο του Μεξικού. Χτες ε, έλαβα, ε, μάλλον μου είπε ο υπεύθυνο της BP ότι λαμβάνουν όλα τα μέτρα για να αποφευθεί η οικολογική καταστροφή. Αυτό μου είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος και βεβαίως η βιομηχανία θα πρέπει να αποτιμήσει την κατάσταση. Μου ε, ανέφεραν ότι ε, λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την προστασία των ε, πολιτών και του περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη νομοθεσία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια συνάντηση με τις βαλτικές χώρες η Φιλανδία μίλησε για πιθανές συνέπειες, δηλαδή αν υπάρχει οικολογική, μια παρόμοια οικολογική καταστροφή στη Βαλτική, τι θα κάνουμε. Αυτό μας απασχολεί ήδη. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να δώσουμε μια γρήγορη απάντηση ή ρύθμιση και δεν υπάρχει καμία εγγύηση απόλυτης ασφάλειας όλα εξαρτώνται από τις πρακτικές της βιομηχανίας. Όμως θα προβάλλουμε αλλαγές ιδιαίτερα με βάση τις έρευνες που γίνονται στον κόλπο του Μεξικού. Ερχόμαστε σε επαφή με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και η Έτιγκερ και Ποτόσνικ, οι δύο επίτροποι, ήρθαν σε επαφή με το βιομηχανικό κλάδο και επίσης προβάλλεται και η αρρωγή MIC και μας δόθηκαν κατάλληλες απαντήσεις. Πρόκειται για μια σειρά πρωτοβουλίων που λήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ως προς το τελευταίο σχόλιο του κυρίου Μαώρο θα ήθελα να πω ότι θα συνεργαστούμε με όλα με όλους τους άλλους φορείς και τα θεσμικά όργανα, διότι όπως είπα η Επιτροπή είναι η οικονομική της Ευρώπης, διότι πρόκειται για αρμοδιότητες που έχουν μεταφερθεί από τα κράτη-μέλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους τους θεσμικούς φορείς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και αυτό αφορά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω λοιπόν ότι υπό αυτό το πνεύμα εταιρικής σχέσης μπορούμε να προχωρήσουμε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη που έδειξαν μεγάλη υπομονή και αντοχή. Αυτή την αντοχή χρειαζόμαστε και για τις οικονομίες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι κηρύσω τη λήξη και της συζήτησης και της ε, συνεδρίασης. Επόμενη συνεδρία σε 12 ημέρες 5 Ιουλίου στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ πολύ.